Δευτέρα μεσημέρι. Δυσκολευόμαστε να ξεκινήσουμε γιατί όλοι ταξιδεύουμε το πρωί, αλλά είναι ήδη 3 και 10, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Βλέπω ήδη ε, γνωστά πρόσωπα, γιατί μετά το Κοτονού τα είπαμε στο Στρασβούργο, έχουμε συνδυάσει ήδη αρκετές φορές. Όσους δεν έχω δει ακόμη όμως, θέλω να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά τελευταίο έτος της τρέχουσα θητείας. Δεν μας μένουν και πολλές συνδριάσεις, αλλά έχουμε να ολοκληρώσουμε σημαντική δουλειά μέχρι να ολοκληρωθεί η θητεία αυτή. Παρακαλώσω και τους συντονιστές και τους βουλευτές να παρίστανται λοιπόν. Έχουμε την ημερησία διάταξη, υπάρχουν κάποιες αλλαγές, τις οποίες θα ήθελα να σας αναγγείλω. Το έχω πει και γραπτός για τις τρεις ε, ε της ΑΚΕΤ 119, 7 Φεβρουαρίου αναβάλλεται η ψηφοφορία αυτή, γιατί υπήρχαν πολλές ε, τροπολογίες και δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις. Θα ξεκινήσουν λοιπόν αύριο στις 10 οι ψηφοφορίες και όχι στις 10 παρατέταρτο. Αν θέλετε παρακαλώ να ενημερώσετε τους βουλευτές ή βοηθοί ότι θα ξεκινήσουμε στις 10 και όχι στις 10 παρατέταρτο. Επίσης, αύριο στις 5.30 θα έχουμε μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για να συζητήσουμε τις ε, τροποποιήσεις στην ε, έκθεση το νέο μέσο 5.30 στο γιαν 2 και 2 το τελευταίο δηλαδή μέρος συνεδρίασης υπάρχουν πολλές τροπολογίες ό,τι αφορά αυτό το μέσο και θα μας τα πει ο εισηγητής. Τέλος Φεβρουαρίου θα γίνει ψηφοφορία. Α, πιο ακόμα, πιο αργά ακόμα, 4 Μαρτίου. Άρα θα έχουμε χρόνο για να καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις. Με αυτές τις αλλαγές μπορούμε να δεχθούμε την ε, ημερήσια διάταξη, παρακαλώ. Ανακοινώς πρόεδρου καταρχάς. δύο συνεδριάσεις με επιτροπές, 24 Ιανουαρίου η πρώτη με την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και η συνεδρίαση την Πέμπτη δηλαδή, 9 με 10 και για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ιεμένη. Στο 3G3 έχουμε λάβει ε, πάρα πολύ άσχημες αναφορές από την Ιεμένη και πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Επίσης, την επόμενη εβδομάδα, 29 Ιανουαρίου, θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και την Επιτροπή Εξωτερικών. Σε ό,τι αφορά την ειδική έκθεση του, μάλλον τι ειδικέ εκθέσει ε, του Ελληνικού Συνεδρίου. Πρώτο είναι η διευκόλυνση για του πρόσφυγε στην Τουρκία. Δεύτερο, το καταπίστευμα για την Αφρική. Τρίτο, έκθεση για τη διαφάνεια ε, και τα προγράμματα που εφαρμόζουν οι ΜΚΟ. 3 με 5. 29 Ιανουαρίου τις λεπτομέρειες θα τις πάρετε. Στο 4Q1 θα γίνει η συνεδρίαση. Επίσης έχουμε ένα νέο υπεύθυνο τύπου που θα καλύπτει το κοινοπλευτικό έργο. Τίλιο Μακάντον είναι το όνομα αυτού του νέου press officer. Έχει εργαστεί ε, στην αναπτυξιακή πολιτική. Ο Τίλο πίσω εκεί είναι. Καλώς ήρθατε και συγχαρητήρια για, την, για τον ορισμό σας δεν εργάζονταν για το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ κατά το παρελθόν. Πρέπει να σας ξανά έχουμε συναντήσει. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, σας καλωσορίζω. Σαν εισερχόμενο στο Κοινοβούλιο. Και ε, ενώπιση και των ευρωεκλογών θα μας ε, τα πείτε πολύ καλύτερα και εσείς. Για το σημείο 3, αποφάσεις των συντονιστών, έχετε τα πρακτικά της 20ης Νοεμβρίου στους φακέλους σας. Ό,τι σχόλιο έχετε πριν το τέλος συνεδρίας στην γραμματεία, αλλιώς θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Μετά έχουμε το σημείο 4, ανακοινώσει ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει κάποια ανακοίνωση. Όχι. Έχει άλλα να μας πει. Θα έρθει και ο Επιτρόπος Τηλιανίδης αύριο στην Επιτροπή μας. Θα μας τα πει λοιπόν σε αυτό το χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε τώρα περνάμε στο πρώτο σημείο ουσία τη διάταξη που είναι αριστερό τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε τον πρόεδρο ε, τη ε, ΕΤΕΠΑ, Βέρνερ Χόγερ. Είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων τον Νοέμβριο με τον Κουντούν και και την Μαριέτα Γιάγκερ που είναι εδώ. Είναι οι αναπληρωτές γενικοί διευθυντές της σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση κομισιών ε, για μια πιο αποτελεσματική οικονομική αρχιτεκτονική για επενδύσει, ε, πρώτη και δεύτερη ανακοίνωση νέα ε, Συμμαχία Αφρικής Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσει εργασία. Και ξέρουμε ότι δίνεται στο νέο μέσο για τα εξωτερικά ζητήματα πολύ μεγαλύτερη έμφαση στα επενδυτικά ταμεία. Το FSD να πάει σε ένα νέο επίπεδο, να ανανεωθεί Επίσης, περισσότερες δαπάνες σε τέτοιου είδους ε, διευκολύνσεις, ώστε να προσελκύσουν περισσότερες επενδύσεις ε, για τις χώρες εταίρους με τους οποίους συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής. Επίσης, σχέσεις ε, με τις τράπεζές μας είναι ένα άλλο θέμα. Είναι σημαντικό που είναι εδώ ο κύριος Χόγερ. Εδώ γνωρίζουμε ότι στο Συμβούλιο οι Υπουργοί συζητούν το νέο αυτό εξωτερικό πλαίσιο, τι μορφή θα έχει και ξέρω ότι και εσείς τα συζητάτε. Έχω επαφές και με άτομα από την BERD και άλλες μεγάλες ε, αναπτυξιακές τράπεζες για να δούμε πώς μπορούμε να εργαστούμε στην Ευρώπη και εμείς θέλουμε τα κονδύλια αυτά να έχουν τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο. Κύριε Χόγερ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τιμή και χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας για να συζητήσουμε σημαντικά ζητήματα και χαίρομαι που μπορώ να συμμετέχω στις διαβλέψεις επιτροπή σας, στις ζητήσεις σας. Έχω μιλήσει δύο φορές στην Ολομέλεια, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης ε, και της έκθεσης της Επιτροπής Προπολογισμού και είναι πολύτιμος αυτός ο διάλογος, εστιάζοντας περισσότερο τώρα στα αναπτυξιακά ζητήματα, διότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι Γίνονται τεκτονικές αλλαγές ε, στα γεωπολιτικά, στο γεωπολιτικό προσκήνιο. Και κάποιες φορές αυτό μας διαφεύγει ε, στη ρουτίνα μας, της καθημερινότητας, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Βλέπουμε την Κίνα πώς τοποθετείται σε διάφορες χώρες όπως και ιδιαίτερα στην Αφρικανική Ήπειρο. Βλέπουμε την απομόνωση της Αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας τεράστιες επιπτώσεις για το πολυμερές σύστημα. Που όπως η και είπα, είναι μέλος αυτή η τράπεζα δηλαδή και άρα θα είναι σημαντικές αλήθειες και προκλήσεις για εμάς τους Ευρωπαίους. Και πρέπει να ανταποκριθούμε και γρήγορα στις προκλήσεις αυτές. Αλλιώς κινδυνεύουμε να αποδυναμωθεί η θέση μας Πιστεύω ότι αυτές οι ανταλλαγές απόψεις ε, είναι πολύ σημαντικές γιατί ενισχύουν τις ε, ε, σχέσεις μεταξύ των τραπεζών. Χαίρομαι και, και του Κοινοβουλίου. Χαίρομαι που μας έδωσε τη δυνατότητα η Λίντα Μακάβανη Πρόεδρος να ανταλλάξουμε απόψεις. Μας γνωρίζετε πιο πολύ για τις επενδύσεις μας εντός Ένωσης. Η Επιτροπή σας βέβαια για πάνω από 55 χρόνια ξέρει ότι δραστηριοποιούμαστε τα μάλα και για τη στήριξη της εξωτερικής και αναπτυξής πολιτικής της Ένωσης σε διάφορες χώρες πέραν των στόνων της Ευρώπης με πραγματικό αντίκτυπο και κάτι πολύ σημαντικό λόγω των όλων και λιγότερων πόρων που στη μας με ελάχιστο κόστος προς τον προπολογισμό. Η Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας πρωταγωνιστής ε, για την ε, συγκέντρωση χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα και για την εξέβριση καινοτόμων χρηματοδοτικών λύσεων για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Δεσμευόμαστε σε project εκτό και εντό ένωση. και είμαστε στη μοναδική θέση να έχουμε εμπειρία σε όλες τις περιοχές και σε όλα τα είδη project. Επίσης, μπορούμε να προσφέρουμε ε, εμπειρία. Δραστηριοποιούμεθα σε όλε τι χώρε του πλανήτη και κυρίω στι ε, χώρε Αφρική, Καραϊβική και Ειρηνικού, που γνώριζε πολύ καλή η επιτροπή σα. Όπω ε, ε, έδειξε και η συμμετοχή μα Συμφωνία Κοτονού, είμαστε έμπειροι, έχουμε τα μέσα, τη δέσμευση για να έχουμε αντίκτυπο στις επενδύσεις. Αντίκτυπος είναι μια πολύ σημαντική λέξη σήμερα. Πλέον δεν έχουμε στόχους όγκου, αλλά αντικτύπου. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δέκα δι ήταν χρηματοδότηση παρασχόμε στην Αφρικανική Ήπειρο. Κινητοποίησαμε επενδύσει τη τάξη του 30 δι περίπου. Βελτίωσαν τη διαβίωση των ανθρώπων. Οι επενδύσει αυτέ δημιούργησαν θέσει εργασία στο τοπικό επίπεδο. Χρηματοδοτούν επίση ΜΜΕ, μικροεπιχειρήσει, εστιάζοντα ε, στι Αφρικανέ γυναίκε. Δίνουμε επίση ενδυνάμωση προ του τοπικού επιχειρηματίε για να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Στηρίζουμε την απασχόληση επίσης, τη βιώσιμη ανάπτυξη και συνεργαζόμαστε και με το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για να μειωθούν τα κενά στον τομέα των υποδομών, σε τόμει όπως είναι η ενέργεια, το νερό, οι μεταφορές. Αυτό σημαίνει ότι με τη χρηματοδότησή μα θα μπορέσουμε, για παράδειγμα, να δώσουμε νερό σε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπου στον Παμάκο, στον Μαλί ή να προσφέρουμε ρεύμα ε, σε πολύ φτωχές περιοχές αγροτικές, στην Κάμπια, στη Γουινέα, στο Μαλί, στην Κένια, να είναι πιο αποτελεσματικό το σύστημα υποχέτευση του Φίτζι, παραδείγματο χάρη, να αντιμετωπίσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα ή να εξυγχρονίσουμε το ε, αστικό συγκοινωνιακό σύστημα στο Ντακάρ ε, για να συνεισφέρουμε αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα. Κυρίε και κύριοι, συνεχώ παρακολουθούμε ακολουθούμε, στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στη σχέση της με τους τέρους από τις χώρες ΑΚΕ, σχεδιάζοντας νέα πρόγραμμα όπως και κάποια εργαλεία επιμερισμού κινδύνων, impact finance για project με αναπτυξιακό αντίκτυπο, πράσινα βιώσιμης ανάπτυξης ομόλογα και άλλες καινοτόμες πρωτοβουλίες όπως το Boost Africa, για να ενισχύσουμε νέους επιχειρηματίες. Για αυτά τα ομόλογα, να πω ότι πριν από 11 χρόνια η ΕΤΕΠ ήταν στην προσταφυλακή σε ό,τι αφορά αυτά τα πράσινα ομόλογα. Τότε, όταν ε, με το χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου είπαμε ότι θα το δοκιμάσουμε με αυτά τα πράσινα ομόλογα, υπήρχε τεράστια επιφυλακτικότητα. Διότι φυσικά ε, πιο εύκολο να το λέει κανείς παρά να εκδίδει τελικά τέτοια ομόλογα, να είναι ο, έπειτα υπόλογος και να είναι διαφανής. Δεν παίρνει ε, ένα λευκό χαρτί, το βάφεις, ε, το χρωματίζεις πράσινο και το λες πράσινο ομόλογο. Πρέπει να υπάρχουν κριτήρια. Τι μπορούμε να αποκαλέσουμε πράσινο ομόλογο. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία. Κανείς δεν θα περίμενε τότε ότι η αγορά αυτή τώρα θα είχε αυξηθεί Μιλάμε για εκατοντάδε δισεκατομμύρια εκδο, εκδοθέντων τέτοιων πράσινων ομολόγων. Και μάθαμε από αυτή την εμπειρία. Είχαμε και με το ΓΔ των Ηνωμένων Εθνών συναντήσεις και μου στήθηκε να ελέγξω κατά πόσον αυτή η ιδέα των πράσινων ομολόγων που εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο στόχο επενδυτικό θα μπορούσε να αναπτυχθεί αυτή η ιδέα και για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης διότι ο Γενικός Γραμματέας των Εθνών ήταν της άποψης πως ναι μεν όλοι χάρηκαν με την επιτυχία της απόφασης για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξη, αλλά σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της απόφασης, μόνο με βάση τα χρηματοφορούμενα, είναι κάτι που δεν θα λειτουργήσει. Δεν θα είμαστε ποτέ σε θέση να χρηματοδοτήσουμε, να φτάσουμε ε, ε, να εκπληρώσουμε αυτού του στόχου μόνο με τα χρήματα των φορολογουμένων. Πρέπει να υπάρξει βελτίωση στον ιδιωτικό τομέα και με την ΕΤΕΠ έχουμε δύο άξονε. Δεν χρηματοδοτούμε μόνο κάποιο project. Πάντοτε προσπαθούμε και από τεχνικής πλευράς ε, να ε, έχουμε τη δέωση επιμέλεια και αν είναι οικονομικά βιώσιμο ιδιωτικοί φορείς ενίοτε είναι έτοιμοι και αυτοί να συμμετάσχουν. Έτσι κεντρώνουμε περισσότερα κονδυλία και εταίρους. Το δεύτερο είναι να έχουμε κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι τα πράσινα ομόλογα, αυτά τα νέα ομόλογα για τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Αν θέλουμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, πρέπει να πω για πρώτη φορά, έχουμε αυτά τα ομόλογα βιωσιμότητας ε, και αξιολόγηση τη βιωσιμότητα ε, πάντα στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. 500 εκατομμύρια και εξαντλήθηκαν αμέσως για πρόσκληση στι αναπτυσσόμενε χώρες και θέλουμε να το επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο αυτό το πρόγραμμα. Αυτά τα ομόλογα στο μέλλον θα στηρίζουν προγράμματα στον τομέα της υγείας και της παιδείας. Πρέπει λοιπόν να συγκεντρώσουμε πόρους ε, αλλά από εκεί που υπάρχουν πόροι. Και έχουμε πολλές δυνατότητες με αυτά τα διεθνώς οργανωμένα κονδύλια και ταμεία, στα και άλλα που μπορούν να παράγουν χρήματα για συγκεκριμένους σκοπούς. Αυτά λοιπόν τα sustainability awareness bonds είναι πολύ, πολλά υποσχόμενα και είναι μέτρα τα οποία θα τονώσουν τις επενδύσεις για μια αηφόρο ανάπτυξη διαρκείας και για τις χώρες δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι οι προκλήσεις ε, για την εξωτερική και αναπτυξιακή πολιτική είναι πολύ σημαντικές ε, με αυτή την αβεβαιότητα γύρω από την, ε, το ρόλο των ΗΠΑ, με το ρόλο της Κίνας που είναι όλο και μεγαλύτερος, ιδίως στην Αφρική και έχοντας πόψη και τις απειλές προς το πολυμερές σύστημα. Πολύ περισσότερες από ποτέ και η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει ηγετική στάση και να αντιμετωπίσει τα παγκόσμια ζητήματα. Επίσης, για να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας ε, για τους βιώσιμού στόχους ανάπτυξης, για να αντιμετωπίσουμε την ε, μεταναστευτική πρόκληση και να πετύχουμε περισσότερα με τους λιγότερους δημόσιους πόρους, χρειαζόμαστε να έχουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας, τα κράτη-μέλη, οι δημερείς οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΕΔ, η ΕΤΕΠ, πρέπει να συνεργαστούν και να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Υπάρχουν πολλέ ανεπάρκειε και αδυναμίε σήμερα στο πλαίσιο τη αρχιτεκτονική χρηματοδότηση σήμερα. Απαιτείται μεγαλύτερο συντονισμό, νέα χρηματοδοτικά μέσα, καινοτόμε τραπεζικέ λύσει. Και αυτό ε, μα έκανε να ξεκινήσουμε στην ΕΤΕΠ ένα προβληματισμό για να δούμε αν ε, θα δημιουργηθεί ε, μια ειδική θηγατρική για ε, θέματα ανάπτυξη εντό του ομίλου. Δεν θέλουμε κάτι εντελώ καινούριο, αλλά να σκεντρώσουμε τι δραστηριότητέ μα στον τομέα αυτό στο πλαίσιο αυτή τη θηγατρική. Και ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση που προσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους Εθνικού αναπτυσσιακούς φορείς να συμμετάσχουν ως μέτοχος. Είμαστε έτοιμοι να διευκολύνουμε, να συντονίσουμε τις εξωτερικές επενδύσεις για τους χάρτη πολιτικής. Αυτό αυτός είναι ο επιμερισμός εργασιών μεταξύ των χαρακτών πολιτικής σε φορείς όπως είναι το Κοινοβούλιο, η, το Συμβούλιο, η κομισιον Και απ' την άλλη υπάρχουν αυτοί οι οποίοι υλοποιούν αυτές τις ε, πολιτικές για να δουλέψουν και να αποδώσουν όλα αυτά τα project. Ε, έχουμε κινητοποιηθεί όλες μας οι υπηρεσίες για την ε, δημιουργία μιας αρχιτεκτονικής αναπτυξιακής χρηματοδότησης κατάλληλης για το σκοπό που έχει να υπηρετήσει. Για να είμαστε μεγαλύτερος δωρητής Είχα γράψει πέρυσι στους ε, συγητές για να πω ποιε είναι οι δικέ μα προτάσει για τη νέα πρόταση για το NDC, αυτό το νέο εξωτερικό πλαίσιο επενδύσεων. Και σίγουρα οι δικέ σα διαβουλεύσει και διαπραγματεύσει για αυτόν τον κανονισμό θα καθορίσει το κατά πόσο η θα μπορέσει να συνεχίσει τις, ε, δράση, τη δράση σε τρίτε χώρε και σε αφρικανικέ και το κατά πόσο επίση θα μπορούν να βελτιστοποιήσουν το δυναμικό της ε, ΕΤΕΠ οι νομοθέτες. Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για το NDICI, τρεις είναι οι βασικές μας αρχές. Να κοδόμψουμε πάνω σε αυτά που αποδίδουν. Δεύτερον, να εξασφαλίσουμε σαφή επιμεσμό εργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων τη Ένωση. Και τρίτον, να βαθύνουμε τι ευρωπαϊκέ εταιρικέ σχέσει. Η αιτήσια έκθεση του Κοινοβουλίου για τι δραστηριότητε τη ΕΤΕΠ εγκρίθηκε την εβδομάδα και υπάρχουν και κάποιες βασικές τροπολογίες στη σχέδιο έκθεσης για το NDC το Δεκέμβριο που δείχνουν και τα δύο αυτά ε, μεγάλη υποστήριξη για έναν ισχυρό ρόλο για την ΕΤΕΠ και ήδη το Κοινοβούλιο ζητεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να διατηρήσει τι φυστάμενε δραστηριότητε στο μέσο εξωτερική πολιτικής μέσω τη εντολή για εξωτερική δανειοδότηση και το ACPIF και είναι σημαντικό κεντρικό ρόλο τη ΕΤΕΠ, που είναι ε, το χρηματοοικονομικό σκέλος τη Ένωση, να αντικατοπτρίζει και, και στη στρατηγική χρηματοδότηση εκτός Ένωση μετά το 2020. Θα δούμε τι θα γίνει με τις τροπολογίες ε, για το NDCI που είναι αύριο ε, στην μεσηδιάταξη της Επιτροπής σας, ολοκληρώνοντας μία έκκληση. Αν θέλετε να έχουμε συγκεκριμένη νομοθεσία θα πρέπει στις ε, τροπολογίες ε, για το τελικό NDCI που θα εγκριθεί 26 ώρες να περιλαμβάνουν τα εξή. Πρώτον, να έχουμε ειδική εντολή για το δημόσιο τομέα για το ΕΤΕΠΑ. Διότι αλλιώς θα χάσει την επαφή που έχει για την ε, δανειοδότηση εκτός των συνόρων. Έπειτα πρέπει να διατηρηθεί η διευκόλυνση επενδύσεων ΑΚΕ 20 δις ιδιωτικών ε, επενδύσεων, μάλλον πίσω του ιδιωτικού τομέα στην Αφρική, μπορούν να υποστηριχθούν χάρη σε αυτό το μέσο, χωρί να υπάρχει κόστο για τον προβλησμό. Επίση, θα πρέπει να υπάρξουν διατάξει που θα διευκρινίσουν το ρόλο τη ΕΤΕΠ. Υπάρχει συμφωνία επιμερισμού εργασία στο πλαίσιο του InvestEU μεταξύ Κομισιών Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΤΕΠ. Έχουμε σημειώσει πρόοδο ως προς το InvestEU. Είναι κάτι που με ικανοποιεί ιδιαίτερα και νομίζω ότι αυτό το προηγούμενο μπορεί να εφαρμοστεί και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον κανονισμό ένδυση. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά ε, το πλαίσιο για το InvestEU. Και θα πρέπει να δούμε και αργότερα ε, πώς θα καταλήξουμε με το NDC. Αυτά, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω στη συζήτηση. Έχω μαζί μου και εμπειρογνώμονες, ε, τη Μαρία Σουπαραγκάν, που είναι αναπληρώτερη γενική διευθυντήρια για τις ε, Και θα με βοηθήσει να απαντήσω στα ερωτήματά σας και στα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Χόγια. Έχουμε έναν από τους συνεισηγητές μας, τον κύριο Γκάλερ, ε, ο οποίος ε, είναι εδώ. Τον κύριο Γκάλερ, συγγνώμη, ο οποίος θα μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω εγώ, αλλά βεβαίως θα πρέπει να με σταματήσετε, γιατί εγώ έχω ένα σωρό ερωτήσεις να υποβάλω στον ομιλητή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, είναι μέρος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως πρέπει να συμμορφώνεται στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα της πράγμα εξαιρετικά σημαντικό για τη δική μας Επιτροπή η οποία δρά και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Υπάρχει ένα πρόβλημα από ό,τι φαίνεται με τη γερμανική διερμηνία κάποιο κουμπί δεν είχε πατηθεί σωστά προφανώς λέει η πρόεδρο. Συνεχίστε κύριε Γέραντς. Ε, να τα πω σε δύο λόγια για να τα καταλάβει και η Μαρία που δεν άκουσε τη διερμηνία. Είπα ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της ενώσεως. Από αυτή την άποψη λοιπόν ε, είναι μέρος της οικογένειας. Εγώ δεν θα ήθελα να φύγετε ε, χωρίς να μας αποσαφηνίσετε λίγο ε, τις ε, δυνατότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και σας εξηγώ τι θέλω να πω. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία χώρα αναπτυσσόμενη που μπορεί να επιτύχει ευημερία χωρίς να περάσει, χωρίς να διανύσει μια φάση βιομηχανοποίησης. Όλες οι χώρες, ίσως με εξαίρεση τη Νέα Ζηλανδία, πέρασαν από αυτή τη φάση. Γνωρίζουμε τις ανάγκες της Αφρικής. Ξέρουμε επίσης ότι σε μερικές χώρες μπορεί να λειτουργήσει καλά το σύστημα. Και ας πούμε, ακούστηκε στην επίσκεψη του Λουξεμβούργου ότι ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι παρόντα στη Ρουάντα και στην Κάνα σε λίγο, σε μερικά χρόνια. Επομένως υπάρχουν χώρες με δυνατότητες, ε, χώρες οι οποίες έχουν ε, ικανό βαθμό διακυβέρνησης έτσι ώστε να προωθηθούν τέτοιου είδους προγράμματα και ε, στοιχεία. Ερώτηση λοιπόν, εάν περιοριστούμε στην ανάπτυξη εκεί που αυτή η ανάπτυξη βρίσκει γόνιμο έδαφος, τότε θα παραμελήσουμε την μισή Ήπειρο της Αφρικής. Παλιότερα ε, υπήρχαν πολλοί οι οποίοι συνηγορούσαν υπέρ δημιουργία συγκεκριμένων ζωνών. Ας πούμε, έχετε μια χώρα με μεγάλη διαφορά, με κανένα βαθμό διακυβέρνησης που δεν μπορεί να γίνει τίποτα ε, και υφίσταται κυρώσεις, ε, Τιμωρείται κατά κάποιο τρόπο ο πληθυσμό, ο κόσμος, λόγω αυτού. Πρέπει να δούμε αν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ζώνη εντός της ε, οποίας ε, και με την συνένεση της κυβέρνησης θα μπορούσαν ε, να δημιουργηθούν κάποιες συνθήκες διακυβέρνησης σωστής, όπου οι επιχειρήσεις θα πλήρωναν φόρους, όπου θα μπορούσε να υπάρξει κατανομή πόρων σύμφωνα με τους χώρους σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό είναι απολύτως... Ε, ε, ε, αυτό μπορεί να γίνει ή όχι. Γιατί εάν δεν ανοίξουμε νέους ορίζοντες, τότε διαγράφουμε το μεγαλύτερο μέρος της Αφρικανικής Υπήρου. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολλούς υπολογισμούς και μπορεί να υπάρξει ε, μία συνεργασία η οποία μπορεί να προσθεθεί στην παραδοσιακή μας συνεργασία αποδίδοντας ένα 7-8-9% ε, και συμβάλλοντας στο μέτρο του δυνατού στη δημιουργία μιας καλής διακυβέρνησης ε, που θα μπορούσε να ε, προσεγγίσει να, κατά κάποιο τρόπο, να προσωμιάσει κατά κάποιο τρόπο με τη δικιά μας. Ε, ξέρετε ότι η Κίνα έχει βάλει το χέρι της παντού και στην αφρικανική οικονομία. Άρα δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια και νομίζω ότι μαζί με την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα έπρεπε να δούμε τι θα μπορούσαμε ε, να κάνουμε στο επόμενο NSI. E Γιατί, ας πούμε, οι αποφάσεις ε, ε, για την, ή τα κονδύλια για την βιομηχανία θα μπορούσαν να προσθεθούν στις διαδικασίες και τα κονδύλια για την ανάπτυξη. Ε, θα μπορούσαν να προσθεθούν στα κονδύλια που δίνονται για την υγεία, για τα σχολεία κλπ. Έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά επειδή θα ξαναπάρω το λόγο αργότερα, να δοθεί δυνατότητα και σε άλλους συναδέλφους. Ε, βεβαίως εσείς ε, πάντα είστε πολύ ευγενείς ε, και ε, διπλωμάτης. Έχουμε έναν πίνακα της ε, Κομισιόν για ένα νέο EFSD. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, μάλλον αυτή η αίσθηση που έχω είναι ότι δεν σας αρέσει η πρόταση της Κομισιόν. Μπορείτε να εξηγήσετε λίγο περί τίνος πρόκειται πραγματικά και τι, ποια είναι, ποιο είναι το διακύβευμα μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Έχουμε μια πρόταση λοιπόν που έχει υποβληθεί. Τι αρέσει, τι δεν αρέσει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Γιατί συζητούν το θέμα και οι υπουργοί. Ε, υπάρχουν κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις που γίνονται. Και βεβαίως ε, θα μας πείτε και αυτά που σας ρωτάω εγώ, αλλά και αυτά που ανέφερε ο, ο Σάρλ προηγουμένως. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν περί τίνος πρόκειται πραγματικά, τι διακυβεύεται εδώ, τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις πρώτες ερωτήσεις. Η μία είναι πολύ συγκεκριμένη, η άλλη όμως ε, ε, γενική αλλά και θεμελιώδης. Εμείς πιστεύω ότι σε μερικές μέρες θα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δείξει ότι μπορούμε να επιτύχουμε συμβιβασμό ή εν πάση περιπτώσει μια καλή κοινή λύση. Και θα, το, θα έχουμε τη δυνατότητα, θα έχετε και εσείς τη δυνατότητα να το πείτε όταν θα φτάσει ενώπιόν σας ε, το, η πρόταση της Κομισιόν. Η συζήτηση που έλαβε χώρα ήταν απαραίτητη έτσι ώστε, όπως είπε και ο Σαλ Γκιόρενς προηγουμένως, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι η διαφορά ανάμεσα ε, στην Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία ή όργανα είναι ότι εμείς ε, είμαστε με, αποτελούμε μέρος του θεσμικού οικοδομήματος. Εμείς είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς είμαστε εσείς και επομένως η διαμόρφωση πολιτικής, η υλοποίηση πολιτικών και στρατηγικών ε, όσον αφορά αυτό το σκέλος των ε, ε, χρηματοπιστωτικών τραπεζικών υπηρεσιών συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο θεσμικό πλαίσιο του NCIDI. όπου ε, μπορεί να, να πρέπει να ληφθούν απαντή, να αποφάσεις με γνώμονα το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιστάσεις όπου ε, όλοι δεν είναι, όλες οι χώρες δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στρατηγικές ανάπτυξης ε, βεβαίως πρέπει να συζητώνται, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι στρατηγικές προκλήσεις σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο ε, κόσμο είναι ότι ε, ε, γύρω από ένα τραπέζι μπορεί να καθίσουν μη Ευρωπαίοι και να συζητήσουν για πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν επίδραση στην ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Έχουμε προγράμματα, το Boost Africa που θέλει να δημιουργήσει ε, νέα προγράμματα για, τις, ε, για την νεολαία της Αφρικανικής ε, Υπήρου Ε, επίσης ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η Παγκόσμια Τράπεζα είναι τέρος μας. Ε, δεν είναι θέμα εάν θέλουμε να συνεργαστούμε ή όχι. Το ζήτημα είναι και ο, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να τεθεί είναι ότι εμείς είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς είμαστε εσείς και σαν τέτοιοι θα πρέπει να διαπραγματευόμαστε και να συμμετέχουμε στην συγχρηματοδότηση κάποιων projects με άλλους εταίρους που έχουν πρόσβαση στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς πρέπει να επιμείνουμε ε, ε, ότι οι κανόνες ε, που θα εφαρμόζονται θα είναι ίδιοι για αυτοί που κανόνες που αφορούν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα, θα διέπουν και τα μη όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δεσμευόμαστε από τους ευρωπαϊκούς ενωσιακούς κανονισμούς και ε, εάν όλοι δεν έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις πρόσβασης και λειτουργίας, τότε δεν δημιουργούνται ίσοι όροι ανταγωνισμού. Και επομένως έτσι απαντώ στη γενική σας ερώτηση. Θα πρέπει να ε, σεβαστούμε τους ρόλους που έχει ο καθένας στην ευρωπαϊκή οικογένεια και να μην ε, θέτουμε ε, όρους που θα αφορούν μονάχα την πολιτική σφαίρα, αλλά θα πρέπει να βρούμε και συγκεκριμένους τρόπους και όπως είπε και ο πρόεδρος Γιούγκερ, όταν ε, συζητούσαμε σε συνέντευξη τύπου ε, την επιτυχία του προγράμματος ε, Juncker, τότε είχε πει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να οργανώσουμε μια εξαιρετικά αρμονική συνεργασία. Μόνο έτσι θα μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Θα μπορούσα να μπω και σε λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος τώρα, γιατί αυτή είναι η κεντρική αρχή. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ είπα ότι θα πρέπει να διδαχτούμε όσο γίνεται περισσότερο από προηγούμενες δραστηριότητες. Ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να μεταφέρουμε αυτούσιο και το πνεύμα το οποίο μας έχει οδηγήσει και εμάς και εσάς στην ε, ε, νέα συνεργασία, το NCIDI. Και επίσης ε, να σας πω ε, ότι είχαμε στην Αντισαμπέμπα τις ε, Africa Days, τις μέρες Αφρικής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ακριβώς εκεί αναφερθήκαμε σε βιομηχανικές ζώνες στην Αιθιοπία. Παρεπιπτόντως δεν να σας πω ότι δίνονται, υπάρχουν προγράμματα που δίνουν συγκεκριμένες δυνατότητες, ευκαιρίες εργασίας σε μετανάστες και αυτό αποτελεί τμήμα της συνεργασίας με την ε, κυβέρνηση της Αντισαμπέμπα. Πιστεύω ότι αυτά τα προγράμματα απασχόλησης ε, μεταναστών κλπ. μπορεί να διευρυνθούν και ε, να δημιουργηθούν υποδομές έτσι ώστε να αυξηθούν αυτές οι δραστηριότητες. Υπάρχει και ένα εκπληκτικό παράδειγμα το οποίο καταδεικνύει ακριβώς ε, την ε, δυνατότητα ανάπτυξης στο Καμερούν ας πούμε όπου σε μια περιφέρεια που ζουν περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι ε, θεσμοθετήθηκε ένα πάρα πολύ απλό ε, σύστημα όπου στα ε, κεντρικά φανάρια στους... Ε, for micro, for, for, for ε, telecommunication. And within very, very short time we have found that... Έχουν τοποθετηθεί κάποια ηλιακά πάνελ για δημιουργία ενέργειας και τώρα επίσης υπάρχει και η δυνατότητα μεταξύ ε, ε, ε, Καμερούν και Γκάνας υπάρχει η δυνατότητα να, να συνεννοούνται και μέσω smartphones σε μια περιοχή η οποία δεν έχει καμία υποδομή ηλεκτρικού. Επίσης, Επίσης, ε, πρόσβαση ε, μέσω κινητών σε λογαριασμούς, σε τραπεζικές υπηρεσίες κλπ. Αυτό είναι ε, το σημαντικό για την Αφρική. Έτσι θα προχωρήσει η Αφρική και η χρήση προχωρημένων τεχνολογικών ή βιομηχανικών ζωνών είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα, κάτι το οποίο συχνά παραβλέπουμε. Εάν δημιουργηθεί ας πούμε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με εφαρμογές τραπεζικές και λοιπές, Οπωσδήποτε θα πρέπει για αυτές τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει λέω να υπάρχει ένα θεσμικό ρυθμιστικό πλαίσιο γιατί διαφορετικά ε, θα δημιουργηθεί ένας παράδεισος για μία ε, εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ενώ ε, δεν θα υπάρχει δυνατότητα για κάποιον άλλο παίχτη. Με τους χρηματοδοτικούς μας εταίρους αλλά και με τους ρυθμιστές, ρυθμιστικές αρχές, θα πρέπει να ε, ε, ε, δώσουμε μια πραγματική τεχνική, αναπτυξιακή αρρωγή, μια πραγματική βοήθεια. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ιδέες οι οποίες θα πρέπει να προωθηθούν και να διευρυνθούν. Αυτά. Ευχαριστώ κύριε Σαρτζεντίνη. Έχει το λόγο ναι, τώρα που ήταν σαφής ε, ο πρόεδρος του CIB, ε, νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να τα πούμε λίγο τα πράγματα κάπως πιο μετριασμένα. Ε, Βεβαίω, οι ίσε ευκαιρίε εξαρτώνται από το που βρίσκεται κανεί ε, στο πεδίο των ίσων ευκαιριών. Αυτοί που εκπροσωπούν λοιπόν μια τράπεζα αναπτυξιακή, εμεί έχουμε στη χώρα μα μια λοιπόν, αναπτυξιακή τράπεζα που θα ήθελα να συνεργαστεί, δεν είμαι εδώ εκπροσωπώντα στην Ολλανδική κυβέρνηση, αλλά όσοι βρίσκονται στον τομέα τη ανάπτυξη και εργάζονται σε μια αναπτυξιακή τράπεζα, θεωρούν ότι είναι κάπω διαφορετικά τα πράγματα στον αφορά το πεδίο ευκαιριών. Επίση, όταν λέτε ότι είναι χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων και πρέπει να τα δαπανίσουν ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δεν ισχύει αυτό στον τομέα της ανάπτυξης. Ε, αναγκαστικά ξοδεύουμε χρήματα μέσω αναπτυξιακών ΜΚΟ ή μέσω οργανώσεων των ΗΕ εθνών και αυτά από τον Ευρωπαίο Φορολογούμενο προέρχονται τα χρήματα. Το να τα δαπανούμε μόνο μέσω ενό Ευρωπαϊκού Θεσμικού Οργάνου δεν είναι ο κανόνα στο συγκεκριμένο τομέα. Καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που λέτε για την ε, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αλλά θυμάμαι εδώ μια συζήτηση δύσκολη όταν δημιουργήσαμε το EFSD και το Κοινοβούλιο επέμεινε ότι θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και θα πρέπει να χρηματοδοτήσει δηλαδή project που άλλες τράπεζες ενδεχομένω να μην θέλουν να χρηματοδοτήσουν επειδή δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει στη συνέχεια επιστροφή των χρημάτων αυτών και υπάρχουν και άλλοι που μπορούν να το κάνουν αυτό και θα ήταν εξαιρετικά υγιές από πλευράς ε, Κομισιών και Κοινοβουλίου να παρακολουθούμε όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους και να τους χρησιμοποιούμε όταν ε, μπορούμε για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή επιτυχή συνεργασία για την ανάπτυξη. Ε, έπρεπε νομίζω να μετριάσουμε κάπως αυτό που ελεγχθεί νωρίτερα. Ναι, να προσθέσω κι εγώ κάτι. Το νόημα της εγγύησης η FSD αφορούσε ακριβώς χώρες που δεν μπορούν να, έχουν πρόσβαση στη δανειοδότηση ε, με τους συμβατικούς τρόπους. Πολύ φτωχές χώρες. Δεν είναι όπως η εσωτερική χρηματοδότηση, δηλαδή, όπου χρηματοδοτούμε ε, για επενδύσεις οι οποίες είναι ασφαλείς επενδύσεις και θα υπάρξει κάποιο αντίκρισμα οικονομικό. Είναι διαφορετικό να εργάζεται κανείς στην Κεντρική Αφρική ή σε κάποιες από τις χώρες αυτές σκεφτήκατε ε, πώς θα διαχειριστείτε τον κίνδυνο, το ρίσκο, θα αλλάξετε μοντέλο και το ερώτημα της Τζούντι ότι πολλά χρήματα διαπανώνται τα χρήματα για την ανάπτυξη από τρίτους. Έτσι, έτσι φτάνουμε και στην ανάπτυξη. Οι άνθρωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν δεν είναι αυτοί οι οποίοι τρέχουν τα προγράμματα, οι ίδιοι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ακούστε, εννοείται ότι χρειαζόμαστε μη ευρωπαϊκούς θεσμούς για να πετύχουμε τους ε, στόχους που έχουμε θέσει. Το... Η Ευρωπαϊκή Ένωση το κάνει αυτό και τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πολλοί και διάφοροι εταίροι με τους οποίους ε, συνεργαζόμαστε, αλλά από την άλλη λογοδοτούμε στους φορολογουμενούς μας. Πρέπει δηλαδή να εξασφαλίσουμε ε, ότι γίνεται σωστή χρήση των χρημάτων αυτών. Ότι ακολουθεί τα πρότυπα τα ευρωπαϊκά. Και αυτό το απαιτούμε από όλους και από όλου του άλλου θεσμού. Και συνεργαζόμαστε συνήθω πολύ καλά με, αυτές τις, ε, με αυτού του θεσμού και δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα το να φτάσουμε στα αποτελέσματα που θέλουμε. Η χώρα σα είναι ο πιο ισχυρό μα σύμμαχο στη χρηματοδότηση, παραδείγματο χάρη. Και γνωρίζουμε ότι τα προγράμματα ανάπτυξη στη Ζάμπια, α πούμε, είναι κάτι διαφορετικό από ένα ζήτημα υποδομών στην Ουαλία. Έτσι είναι τα πράγματα. Όμω, παρόλα αυτά πρέπει να κινηθούμε επαγγελματικά και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα πρότυπα αυτά τα επαγγελματικά θα γίνουν σεβαστά και εκεί. Διαφορετικά μπορεί να μην φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε. Υπάρχει βεβαίως μια μεγάλη διαφορά μεταξύ ενός ε, δωρη, μιας, ε, μιας, ε, θεσμού που παίζει το ρόλο του δωρητή και μια δανειοδοτική οργάνωση, δεν μπορούμε εμείς να δίσουμε, να δώσουμε υποτροφίες. Εμείς δίνουμε ένα δάνειο και το οποίο πρέπει να πληρωθεί. Δηλαδή κάποτε πρέπει να πάρουμε πίσω τα χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, δεν είναι να κεφαλοποιήσει τα χρήματα των φορολογουμένων. Είναι να χρηματοδοτήσει project με 62-90 δις ε, έως και 90 δις το χρόνο και για να το κάνουμε αυτό δανειζόμαστε χρήματα στις αγορές. Κάποιοι περήφανα λένε ότι είμαστε πιο μεγάλη πολυμερής ε, χρηματοπιστωτική οργάνωση, αλλά από την άλλη είμαστε και από τους μεγαλύτερους ε, ε από τις κεφαλαίες Γιατί να μας θα δώσουν τα χρήματα αυτά. Ξέρουν ότι έχουμε τεχνική πραγματονομοσύνη για να πούμε ότι ένα project είναι καλό και ότι έχει νόημα από οικονομικής πλευράς. Να πω λοιπόν ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα project, σε, μια δύσκολη, σε ένα δύσκολο περιβάλλον στην Αφρική από ένα project ε, στο κέντρο του Μονάχου. Πάντα όμω, σε όλε τι περιπτώσει πρέπει να είμαστε επαγγελματικοί, επαγγελματίε στην προσέγγιση μα. Ναι, ναι, είστε πεπισμένοι εσεί για την επαγγελματικότητά σα όμω οπότε λογικά δεν θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα. Ναι, βεβαίω και είμαι πεπισμένο για την επαγγελματικότητα, αλλά για να είμαι ακόμα πιο αξιόπιστο, θα δώσω το λόγο στην συνάδελφο εδώ, που, είναι η πιο επαγγελματία. Ακούστε, ήθελα να διευκρινίσω ότι εμεί δεν είμαστε κατά τη ανοιχτή αρχιτεκτονική, για να είμαι σαφή, έτσι, τη ανοιχτή δομή. Απλώ τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και συμμετέχουν και τα διμερεί όργανα και τα μη ευρωπαϊκά. Να το συζητήσουμε. Επίσης, τα διμερεί προγράμματα χρηματοδοτούνται από εθνικά ε, εθνικές κυβερνήσεις, τη γερμανική, την ολλανδική, τη γαλλική, εξαρτώνται από, από εκεί. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Μεδίσεων έχει χρήματα από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Γι' αυτό λοιπόν η συζήτηση που έχουμε, για να έχουμε μια βάση, ε, να, να μπορούμε να βασιζόμαστε δηλαδή σε κάποια ε, χρήματα και σε κάποιες δραστηριότητε προβλέψιμες για να μπορούμε να συντηρήσουμε τις εργασίες μας. Και αυτό λέμε. Δεν λέμε να συμμετάσχει μόνο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει θέση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν υπάρχει αναγνώριση της ειδική φύσης ε, αυτής, αυτής της τράπεζας. Δεν θέλουμε λοιπόν να, να αποκλείσουμε άλλου. Θέλουμε να υπάρχει μια βάση που να επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συμμετάσχει μαζί με άλλου. Διότι οι προκλήσει είναι μεγάλε και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτό θα γίνει με βάση τον ευρωπαϊκό τρόπο και τι ευρωπαϊκέ αξίε. Ε, εκεί, εκεί έχει νόημα η συζήτηση. Δεν υπάρχει πιο αποτελεσματικό εργαλείο από την εντολή εξωτερικής ε, συνεργασίας. Γι' αυτό και πρέπει να συνεχιστεί. Ε, τώρα, υπάρχει το θέμα της διευκόλυνσης ε, επένδυσης. Ε, να μην πετάμε αυτά που λειτουργούν. Έγινε και ένα σχόλιο για το σχέδιο εξωτερικής, εξωτερικών επενδύσεων αποφασίστηκε να κάνουμε κάτι που δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Είναι ήδη πολλά αυτά που κάνουμε. Έγινε μια συζήτηση για την κεντροαφρικανική δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Έτσι, αν υπάρχει μια έθρα στη χώρα είναι αυτή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εξετάζουμε ένα project κινητή τηλεφωνία, όπω αυτό που παρουσίασε ο πρόεδρο προηγουμένω και το οποίο εφαρμόσουμε ήδη στο Καμερούν και αλλού. Θέλουμε να, να προσθέσουμε ένα τέτοιο σύστημα στην κεντροαφρικανική ε, δημοκρατία. Ως, θα συμμετάσχει ο ιδιωτικό τομέα, ορισμένε φορέ ο ιδιωτικό τομέα είναι πιο εύκολο ε, στη συνεργασία προ το δημόσιο, για να δούμε πώ μπορούμε να έχουμε πρόσβαση ε, στι πιο απομακρυσμένε περιοχέ, ε, στην Ήπεθρο. Και βεβαίω πρέπει να συνεργαστούμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα το κάνουμε μόνοι μα. Και με την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία εκεί και με την ε, ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λοιπόν έχει ήδη τα εργαλεία και πρέπει να τα χρησιμοποιήσει για να φέρει αποτελέσματα ακόμα και σε αυτέ τι έθραυστε χώρε. Έχουμε κάποια αντίγραφα, μπορούμε να σα δείξουμε και άλλα παραδειγμάτων επιχειρήσεων σε αυτέ τι χώρε. Ε, κάποιοι λένε ότι εμεί ασχολούμαστε μόνο με μεγάλε υποδομέ, ότι λειτουργούμε μόνο, μόνο στο δικό μα περιβάλλον. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Μπορούμε να κάνουμε και ε, ε, σχέδια υψηλού κινδύνου ε, σε άλλα περιβάλλοντα ε, με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Αυτό δεν το ξέρετε. Μεγάλα τα ποσοστά συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Α αφήσετε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να έχει μια βάση και μετά συνεργαστούμε όλοι μαζί. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε όλο τον κόσμο. Η πρόκληση είναι τεράστια η SDG του 2030 δεν είναι μακριά. Ε, οπότε πρέπει να προχωρήσουμε. Είναι εδώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, ο Νόελ θέλει να ζητήσει κάτι πρώτα. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποιες παρατηρήσεις και καμία-δυο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι υπάρχει αυτή η υποχρέωση λογοδοσία είναι φυσιολογικό αυτό και θα πρέπει να τηρούνται τα πρότυπα, αλλά βασικά εγώ θεωρώ ότι σε ό,τι αφορά τι πρωτοβουλίες των τραπεζών θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο για την ε, ε Κομισιόν, γιατί εμεί έχουμε στη Γερμανία ε, εμπειρία που βλέπουμε πού είμαστε επιτυχείς και πού δεν είμαστε είναι ένα πολύ σημαντικό κριτήριο που δεν θα πρέπει να το παραβλέπουμε. Σε ό,τι αφορά τα βασικά σημεία τα οποία ανέφερε ο πρόεδρος της συμφωνώ να στηρίξουμε ε, προγράμματα με έμφαση στις γυναίκες, υλοποίηση των ε, βιώσιμων στόχων ανάπτυξης. Φυσικά και αυτά πρέπει να υποστηριχθούν. Τώρα, δύο ερωτήσεις σε ό,τι αφορά αυτό το Sustainable Awareness Bond και το Subsidiarity Group. Μάλλον τη θηγατρική εννοεί ο μιλητής, ε, τη θηγατρική αυτή. Πώς τα βλέπετε. πώς μπορούν αυτά να συνδυαστούν με κάτι που ανέφερε και η πρόεδρος. Υπάρχουν έφραυστα κράτη Αφρικανική Δημοκρατία, Κονγκό, Μαλή, Τσάντ. Εκεί και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι έτοιμη η ΕΤΕΠ να πλαισιώσει επενδύσεις ψηλού κινδύνου. Και σε ό,τι αφορά και τη Αφρικανική Επενδυτική Τράπεζα και τις σχετικές άλλες ε, τράπεζες υπάρχει καλή συνεργασία. Αυτή η τράπεζα είναι έτοιμη, η Αφρικανική Επενδυτική Τράπεζα, να αναλάβει επενδύσεις ψηλού Καλό θα ήταν, πολύ καλό, δηλαδή ε, και οι δύο ομόλογοι, Ευρωπαϊκή και Αφρικανική Τράπεζα, να αναλάβουν επενδύσεις ψηλού Και το τελευταίο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά συνολικά και στην ευρωπαϊκή πολιτική νομίζω ότι πλέον είμαστε εστιασμένοι στην Αφρική, πολύ πιο έντονα. Αν δει κανεί ε, τις ε, δαπάνες, ε, είναι το μεγαλύτερο επίκεντρο, ακόμα περισσότερο και από τις χώρες γειτονίας στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν γνωρίζω ακριβώς το ποσοστό, αλλά νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πηγαίνει εκεί και νομίζω λιγότερο, δηλαδή πάνω από το 50 μπορεί να πηγαίνει σε αυτές τις ε, χώρες και γύρω στο 20% σε χώρες ΑΚΕ. Είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε περισσότερο σε εισαναπτυξιωσόμενες χώρες. Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Χόγερ, λέει πρόεδρος, και μετά θα ζητήσω από την Κομισιόν πάρει Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τα Sustainability Awareness Bonds, τα ομόλογα, πρόκειται για μια πρόκληση. Διότι υπάρχουν ε, κονδύλια ε, τα οποία έχουμε ε, για συγκεκριμένους στόχους. Δηλαδή οι επενδυτές θέλουν να ξέρουν, να είναι βέβαιοι ότι θα πάνε στο στόχο τα χρήματα και δεν θα εξαφανιστούν στα ταμεία της ΕΤΕΠ γενικά. Πρέπει δηλαδή να οριστεί συγκεκριμένα το εκάστοτε project και το ομόλογο. Με τα πράσινα ομόλογα έχουμε τη σχετική εμπειρία. τη διαπρόκληση είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτά τα ομόλογα έπρεπε ε, να οριστούν με βάση διεθνή συμφωνία. Και τώρα θέλουμε να το βελτιώσουμε το σύστημα αυτό, γιατί πολλές φορές υπάρχουν κάποια project από διάφορους θεσμούς που παίρνουν την ετικέτα πράσινο, αλλά τελικά τι πράσινο έχουν, ε, διαρωτώ με ορισμένε φορέ. Ε, χρειάζονται κριτήρια λοιπόν. Πολύ συγκεκριμένα. Το ίδιο ισχύει και για τα δεύτερα αυτά ομόλογα. Το νερό είναι ο πρώτο τομέα που έχουμε επιλέξει για να στηρίξουμε την πρόταση των Ηνωμένου Επειδή μπορούμε να έχουμε κάποια συγκεκριμένα project και να κάνουμε και ένα χαρτοφυλάκι διαχείριση κινδύνου. Το νερό είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Ένα άλλο τομέα είναι η παιδεία και η υγεία τα επόμενα κάνα δύο χρόνια. Πρόκληση πάντω μεγάλη είναι διότι απαιτεί τεράστια συνεργασία επιτόπου. Και είναι και πολύ δύσκολο να καταλήξει κανεί σε παγκόσμια συμφωνία. Αυτό καταδεικνύεται και από την πρόκληση που αντιμετωπίσαμε στο πλαίσιο χάρη τη ομάδα των 20, του G20 σε άλλα φόρματ. Για, να... για το asset class, ό,τι αφορά τα... τις υποδομές. Γιατί είναι δύσκολο να προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις. Ξεκίνησε πέντε χρόνια πριν η συζήτηση αυτή και ακόμη δεν έχουμε καταλήξει συμφωνία. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη μια ταξινόμηση ή ταξονομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο ε, και οι Τράπεζε τη Ευρωπαϊκής Ένωση πάντοτε πρέπει να διατηρούν μια ευθραυστή ισορροπία μεταξύ της δραστηριότητα ε, στι γύρω χώρε και της δραστηριότητα ε, στον ευρύτερο κόσμο. Αφήνω στην συνάδελφό μου να απαντήσει, γιατί ίσως έχει στοιχεία στη διάθεσή της. Δεν ξέρω αν υπάρχει ε, αυτή η αντιστοιχεία, αν είναι 80 προς 20. Υπάρχει ευθύνη πάντως ε, για τις χώρες γειτονίας, για τις ενταξιακές υποένταξη χώρες και τα μελλοντικά, τα δυνητικά μελλοντικά μέλη. Τώρα, επανεστίαση σε αμψόμενες χώρες. Αυτό θα ξεπεράσει κατά πολύ τις χώρες ΑΚΕ από στρατηγικής πλευράς. Υπάρχει τεράστια ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη Λατινική Αμερική. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα, αλλά γι' αυτό απαιτείται εντολή. Και η εντολή αυτή δεν μπορεί να έρθει από το ELM ή από αυτή τη διευκόλυνση της επενδύση που μακάρι να την προωθήσουμε περισσότερο, δεν είναι στα δικά μας χέρια όμως. πρέπει να σας πω ότι πολύ καλά κάνουμε και επενδύουμε περισσότερο ή θα έπρεπε να επενδύσουμε περισσότερο στους εταίρους μας ε, αναπτυγμένες χώρες και ανεπτυσσόμενες χώρες, κυρίως αναδυόμενες αγορές. Το λέω από στρατηγικής πλευράς. Έχουμε μια πρόκληση που θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Για να δει κανεί τι γίνεται με την Αφρική, την Κίνα, την Λατινική Αμερική και τη νέα θεώρηση στι ΗΠΑ και το τι κάνει εκεί η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Όλα αυτά μα κάνουν να πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βάση στην εκπροσώπηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον ψώμενο κόσμο και στι αναδεόμενες αγορές τουλάχιστον 10% πρέπει να είναι. Και για τα στοιχεία, τα αριθμητικά σε ό,τι αφορά τις σχέσεις ε, γειτονία, η Μαρία, ναι, Κάποιε πιο συγκεκριμένε ε, εξηγήσει. Ό,τι αφορά την περιφερειακή κατανομή όμως, από ότι αυτό δεν το αποφασίζουμε εμείς, αλλά χάρακτη της πολιτικής. Άρα δεν είναι ε, στα χέρια μας. Εμείς ε, κάνουμε αυτό που μας λένε να κάνουμε στις διάφορε περιοχές. Τι κάναμε. Για την Αφρική συγκεκριμένα, έχουμε αναβαθμίσει τη δραστηριότητά μας τα τελευταία χρόνια Πρόκειται για μια μείζον πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την εσωτερική πολιτική, μιλάει για την κατάσταση στην Αφρική. Και αν δει κανεί και τη δημογραφική εξέλιξη, εάν δεν δράσουμε τώρα, τα πράγματα θα επιδεινωθούν πολύ. Εξού και εστιάζουμε στις προσπάθειε μας, εστιάζουμε πραγματικά στην Αφρική, ω Ήπειρο, ε, Βόρεια Αφρική, αλλά με μεγάλη έμφαση στην Ποσαχάριο Αφρική και πέρυσι το 30% της δράσης μας ε, ήταν στην Αφρική, για να έχετε μια ιδέα. Αλλά μας ζητείτε να κάνουμε πολλά και στις ε, γειτονίε, στις χώρες γειτονία. Αυτό μας το ζητούν οι χαρακτήρες πολιτικής και εκεί ε, εστιάζουμε στις προσπάθειές μας. Λατινική Αμερική, Ασία, το είπε και ο Πρόεδρος. Έχουμε και την κλιματική δράση για τη μείωση των εκπομπών για αυτές τις χώρες. Μιλήσατε και για τις χώρες Καρυβικής και Ειρηνικού. Αναλογικά ε, δρούμε σε ό,τι αφορά την εντολή που έχουν για τις χώρες ΑΚΕ. Προσαρμογή ε, στην κλιματική αλλαγή. Μιλάμε για μικρά νησιωτικά κράτη που είναι πολύ ευάλωτα και στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Άρα θέλουμε να έχουμε ανθεκτικές υποδομές ε, ως αλλαγή του κλίματος και μετριασμό της αλλαγής του κλίματος. Αυτές είναι οι πολιτικές που έχουμε αναλάβει. Είπατε Μαλή, Τσάντ. Ακούστε, σε όλες αυτές τις χώρες προσπαθούμε να έχουμε κάποιες εταιρικέ σχέσεις ε, βέβαια, κυρίως επειδή ξέρουμε τα όρια μας. Για το Τσάντ πρέπει να σας πω ότι συνεργαζόμαστε με τα όργανα του ΟΗΕ που είναι επιτόπου, είναι πιο κοντά στην κυβέρνηση και μπορούν να μας ε, βοηθήσουν και στη μόχλευση, ώστε κάθε ευρώ το οποίο δαπανάτε να έχει το μέγιστο δυνατό επενδυτικό αποτέλεσμα. Εκεί εστιάζουν οι δραστηριότητες μας στην περιοχή. You Μη λησμονείτε ότι η τράπεζα είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία, ας πούμε. Έχουμε 3.500 ε, υπαλλήλους ε, και με ένα ισοζύγιο 600 δις. Ε, αν κάνετε τη σύγκριση λοιπόν με την Παγκόσμια Τράπεζα, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα συνολικό για συνολικά 18.000 ανθρώπους ε, και μονάχα ένα πολύ μικρό ποσοστό έχουμε στο Λονδίνο και επομένως από τη στιγμή που δεν έχουμε το προσωπικό που θα θέλαμε και τους πόρους που θα θέλαμε πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστούμε με άλλες ε, μιλάμε και με την France Development που μας, με, τους οποίους συνεργαζόμαστε όσον αφορά το προσωπικό ε, και με ένα σωρό άλλους οργανισμούς. Ιδιαίτερα βέβαια με την Παγκόσμια Τράπεζα και με την Τράπεζα για την Ανάπτυξη της Αφρικής. Ε, στενή συνεργασία με τους άλλους. Ε, αυτός είναι ο μόνος δρόμος γιατί εμείς θέλουμε να παραμείνουμε ισχυροί. Ορισμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας ε, επικρίνουν γιατί δεν έχουμε και όλα τα γραφεία που θα, πρέπει, που θα έπρεπε να έχουμε. Ε, είναι γεγονός ότι λίγοι δουλεύουν στο Λουξεμβούργο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ, λέει η Πρόεδρος. Να ξεκαθαρίσω όμως και κάποια πράγματα. Η Μεριά Θεγιάγκερ είναι εδώ και η Κομισιόν προτείνει λοιπόν κάποιες αλλαγές για το FSD+. Γιατί τις προτείνει. και στην συζήτηση που θα γίνει ποια θα είναι η κυρίαρχη σκέψη. Γιατί βεβαίω υπάρχουν και χώρε οι οποίε έχουν αναπτυξιακέ τράπεζε, υπάρχουν αυτοί που λένε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, με καλύτερο τρόπο τα χρήματα για τα αναπτυξιακά προγράμματα, γιατί λένε ότι ούτε ή άλλως ε, πληρώνουν οι Γερμανοί, οι φορολογούμενοι, οι Γάλλοι, φορολογούμενοι, οι, Λουξεμβούργοι κτλ. Και εμείς θέλουμε οι δικέ μας αναπτυξιακές τράπεζες να χρησιμοποιούν και να δαπανούν τα χρήματα αυτά και όχι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. και κάθε φορά που γίνεται λόγος για αύξηση του καταπιστεύματος ε, οι χώρες λένε άμα έτσι κι αλλιώς εμείς πληρώνουμε ήδη πολλά. Μήπως η Κομισιόν θα μπορούσε να μας δώσει τα φώτα της ε, γιατί προτείνετε αυτές τις αλλαγές ε, στρατηγικής. Και επίσης κατά τη δική σας άποψη πώς προχωρούν οι συζητήσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε αγαπητή Λίντα να πω εξ ονόματο της Κομισιόν πρώτα απ' όλα ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρο Χόγια για την ε, εξαιρετική παρουσίασή του. Γνωρίζετε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προβλέπεται από τις ε, συνθήκες και έχει συνεργαστεί στενά με την Κομισιόν εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, και είμαι ιδιαίτερο ευτυχή για αυτήν την συνεργασία και τον διάλογο. Αλλά όπως είπε και ο πρόεδρος Χόγια προηγουμένως, εάν θέλουμε ε, να υλοποιήσουμε τους στόχους ε, της βιώσιμης ανάπτυξης ε, οπωσδήποτε χρειαζόμαστε βοήθεια από παντού. Χρειαζόμαστε εταίρους, χρειαζόμαστε πόρους και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και συγκεκριμένες αρχές βάσει των οποίων θα υλοποιήσουμε τα προγράμματα. Συμφωνώ με τον Πρόεδρο ότι χρειάζεται καλύτερη συνεργασία και καλύτερος σωστότερος συντονισμός. Και από την πλευρά μας, ε, από την πλευρά της Κομισιόν, ζητούμε, αυτό που αποζητούμε είναι ο αναπτυξιακός αντίκτυπος και μια νέα χρηματοδοτική αρχιτεκτονική για τα χρήματα που επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα οργανώσουμε ένα σεμινάριο τις 24 ε, του μηνός, ε, το απόγευμα της Πέμπτης δηλαδή, και με μεγάλη χαρά σας προσκαλώ και εσάς. Ε, και στο σεμινάριο αυτό θα ξαναπούμε ότι για την υλοποίηση του EFSD ε, και συγκεκριμένα για τα έξι προγράμματα τα οποία έχουμε για τις ε, ε, πλατφόρμες μεταποιήσεις τις πλατφόρμες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις, τους τίτλους που σχετίζονται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ. Για την υλοποίηση λοιπόν του EFSD μέσω αυτών των έξι πλατφορμών βασιστήκαμε στη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ευελπιστούμε ότι και το θέμα των εγγυήσεων θα κλείσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όσον αφορά την αρχιτεκτονική, να σας πω ότι η Κομισιόν πιστεύει ότι χρειαζόμαστε μια νέα αρχιτεκτονική αν θέλουμε να έχουμε ε, ε, επενδύσεις και σε πιο ευάλωτες χώρες και σε πιο επικίνδυνα απόψη επενδύσεων ε, περιβάλλοντα. Και βασιζόμαστε βεβαίως σε όλους τους εταίρους και κυρίως στους Ευρωπαίους ε, γιατί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι κανόνες βάσει του άρθρου 11 ε, του EFCD, EFSD, συγγνώμη. Μέχρι τώρα εμείς ε, έχουμε δαπανίσει 1,5 ε, δίσε από τις ε, εγγυήσεις. Οι χώρες έχουν δώσει το πράσινο φως και πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι και το πρότυπο επενδύσεων για το μέλλον, ε, δηλαδή ανάπτυξη μέσω στοχευμένων επενδύσεων. Και άλλωστε αναφέρεται και στην έκθεση ότι ε, με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και κάτι τελευταίο για τις μελλοντικέ εγγύσει. Ε, ναι, θα υπάρχει και δυνατότητα ε, δημοσίων, δημοσίου δανεισμού και θα υπάρχει και η δυνατότητα και ιδιωτικού δανεισμού. Ξέρετε ότι για τις νέες εγγύσεις προτείνουμε έξι δις και Οπωσδήποτε μπορούμε να υποστηρίξουμε και τις τροπολογίες της Επιτροπής σας ε, των προϋπολογισμών, γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία και επομένως αποτελεσματικότερο αντίκτυπο. Και δύο τελευταία λόγια. Ναι, policy first. Εμείς θέλουμε ε, να έχουμε συγκεκριμένη στρατηγική και μετά να ακολουθήσει και ο προγραμματισμός και πιστεύω ότι στο μέλλον θα έχουμε και διμερείς ε, συνομιλίες ε, με την ε, τράπεζα που θα επιβεβαιώσουν ότι η τράπεζα παραμένει ο κυριότερος ε, και πιο σημαντικός εταίρος μας ε, όταν μιλάμε για διαχείριση κινδύνου και για ισχυρό αντίκτυπο. Αυτά σας περιμένουμε την Πέμπτη το απόγευμα. Την ε, Παρασκευή θα έχουμε και συζήτηση για τη στρατηγική του EFSD και ευελπιστώ ότι θα σας δω και την Παρασκευή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη διευκρίνηση. Δεν βλέπω να θέλει κάποιο άλλο μέλος ε, τον λόγο, αν θέλει να επανέλθει κάποιο. Έχετε κάποια συμπεράσματα, κύριε Χόιτ, να μας πείτε. Αύριο θα ζητήσουμε τι τροπολογίε μας, ε, θα ψηφίσουμε σε πέντε εβδομάδε περίπου. Ναι, ήταν πραγματικά μια πολύ καλή ευκαιρία να τα πούμε και σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γέγκερ για τα πολύ ε, σαφή λόγια και το πνεύμα συνεργασία, διότι αυτό χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Όλοι γνωρίζουμε ότι θα πάρει πιο πολύ χρόνο από το InvestEU αυτό. Θα έχουμε νέο κοινοβούλιο, νέα κομισιόν. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε κατά νου ότι και το Συμβούλιο, αλλά και το Κοινοβούλιο θεωρώ, αναμένουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσουν να θα μπορέσει να τα βρει μαζί μας, ε, να έχουμε την ίδια φωνή, κοινή φωνή, να μην ασχολούμαστε δηλαδή με τι διαφωνίε μας, αλλά με τις λύσεις που μπορούμε να βρούμε. Θα πάρει χρόνο και είναι σημαντικό μετά από αυτό το δύσκολο κομμάτι με το InvestEU να φτάσουμε σε ένα σύστημα, μια εταιρική σχέση που να μπορέσει να, κάποια στιγμή να περιλαμβάνει και την NDSCI. Ευχαριστώ πολύ για την σαφήνεια και την επιθυμία να βρεθεί μια λύση. Εμείς είμαστε ευρωβουλευτές, ε, υπάρχουν εμπειρογνώμονες, εσείς εμπειρογνώμονες της Κομισιόν. Καλό είναι λοιπόν να βρείτε έναν τρόπο να συνεργαστείτε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο ε, και, την, ε, και τους συνοδούς του. Okay, colleagues. Λοιπόν, όσοι συνάδελφοι αποχωρούν, να σου αποχωρήσουν ησύχως και να περάσουμε στο σημείο 6. Κάποιος από την Κομισιόν θα μας κάνει μια παρουσίαση, ο Φέλιξ από την ΤΕΦΚΟ όχι την υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης όμως, την ΤΕΦΚΟ. Okay, colleagues, move on to item 6 now, which is next... Σημείο 6, λοιπόν, μια ανταλλαγή απόψεων ε, για την κοινή σκευελοντική έκθεση σχετικά με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και την, και την εφαρμογή της ατζέντας του 2030. Είναι μια έκθεση που σχετίζεται με τη Συμφωνία για τη Γενική Συνένεση για την Ανάπτυξη. Εξετάζουμε πώς θα η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη από κοινού αναπτύσσουν πολιτικές για να, εφαρμόσουν τα VSTGs. Είναι σημαντικό αυτό το κείμενο, διότι είναι μέρος αυτών που θα παρουσιάσει στη Νέα Υόρκη αργότερα φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση στην έκθεσή της στο Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την υλοποίηση των STGs. συνεργαζόμαστε και με την Επιτροπή Περιβάλλοντο ε, για να προετοιμάσουμε μια γνωμοδότηση ιδία πρωτοβουλία για το πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει στην εφαρμογή των SDG και εσωτερικά και εξωτερικά. Υπάρχει και ένα εργαστήριο ακρόαση σε δύο εβδομάδε από αυτού με τον Επίτροπο Τίμερμαντ. Θα έρθει και ο Τζέφρι Σάξ ε, ω προσκεκλημένο ομιλητή από τα Ηνωμένα Έθνη Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο για το Κοινοβούλιο με βάση την έκθεσή σας που θα προκύψει ε, τον Απρίλη η έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΦΚΟ και εμείς τώρα θα είμαστε σε προλογική περίοδο γι' αυτό καλέσαμε τον Φέλιξ Φερνάντες Σο να μας πει τι γίνεται έτσι ώστε να έχουμε μια εικόνα του τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτού τι έχει κάνει τα δύο τελευταία χρόνια για να το συμπεριλάβουμε και στην έκθεσή μα, αυτή την κοινή έκθεση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, σε περιπτώσει. Βλέπω ότι η κυρία Θεοχάρο είναι εδώ ή δεν είναι εδώ, αλλά είναι κάποιο που την αντικαθιστά. Ε, μπορείτε να μα πείτε, κύριε Φερνάντε, κάποια λόγια. Είμαστε, ε, εν πάση περιπτώσει, στο, στο δρόμο για το να πετύχουμε το 2030 τους στόχους μας. Έχουμε ξεκινήσει καλά. Ευχαριστώ Λίντα και καλό απόγευμα σε όλους. Ναι, αυτή η έκθεση, η κοινή σκηφολογική έκθεση δεν είναι εύκολο, δεν ήταν εύκολο να προετοιμαστεί. Ξεκινάμε με κάποιες ε, οδηγίες που έχουμε λάβει, θέλουμε ε, μια κοινή έκθεση Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα κράτη-μέλη, οπότε το πρώτο, το η πρώτη επιπλοκή είναι όχι, να καταλάβουμε όχι μόνο τι κάνουν οι Ευρωπαϊκοί Ένωση, αλλά και τι κάνουν και τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την υλοποίηση τη Ατζέντα 2030. Έτσι λοιπόν αυτή η έκθεση, η κοινή συγκεφαλωτική έκθεση, δίνει μια εικόνα του τι κάνουμε εμεί ω δωρητέ πώ εφαρμόζουμε την ατζέντα. Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό, σύμφωνα με, το, με τη συνένεση, με το consensus που πρέπει να προεσιώσουμε μια έκθεση κάθε τέσσερα χρόνια. 2015 λοιπόν συν 4, 2019. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά που από τα κράτη-μέλη, προσπαθούμε να φτάσουμε στη σωστή προσέγγιση. Είμαστε σε αρχική φάση ακόμα, μαθαίνουμε, είμαστε στα δύσκολα. Επίσης προσπαθούμε να βασιστούμε στην το υπάρχον σύστημα αναφορών. Υπάρχουν εκθέσεις, αναφορές στον ΟΣΑΝΤΑ και έχουμε το ΕΙΑΤΗ. Προσπαθούμε να κάνουμε μια περίληψη αυτών που κάνουμε. Λαμβάνοντα υπόψη ότι η Ατζέντα 2030 βέβαια είναι πολύ ευρεία. 17 στόχοι σε τομεί όπου τα κράτη-μέλη και η Ένωση είναι εξαιρετικά δραστήριοι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε κάποιε επιλογέ. Είναι σημαντικό να το ξέρετε αυτό διότι πρέπει να είμαστε και σχετικά συνεκτικοί, πρέπει να κάνουμε κάποιες επιλογές. Έχουμε λοιπόν εδώ μια περίληψη. Θέλουμε να δούμε πρώτα πώς οι Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν αλλάξει τον τρόπο εργασιών τους ε, λόγω της ατζέντα και λόγω της συνένεσης, λόγω του κονσένσους και πώς όλοι έχουμε βελτιώσει ε, την προσέγγιση μας για τα, και την υποστήριξή μας στα, στα τεστ SDGs. Δεν έχει αλλάξει μόνο η φιλοσοφία μας και ο τρόπος εργασίας μας, αλλά και το εύρος των εργασιών. Όλοι μας και τα κράτη-μέλη εργαζόμαστε στα πλαίσια όλων των SDGs. Δεν εργάζονται βέβαια όλα τα κράτη-μέλη πάνω σε όλα τα SDGs, αλλά όλοι μαζί, η Ευρωπαϊκή Ένωση και, η Ευρω... και τα κράτη-μέλη, σημαίνει ότι, όλοι... ότι καλύπτουμε όλο το φάσμα, οπότε είναι περίπλοκο. Τώρα για το περιεχόμενο. Τα βασικά μηνύματα για το τι έχουμε πανεξετάσει, τι έχουμε βελτιώσει, ε, μια νέα πρωτοβουλία, κάποιες νέες πρωτοβουλίες ε, από το 2015 ε, για την ισότητα των δύο φύλων, για την ε, αστική ανάπτυξη, τη σχέση ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, διατροφή, ε, διατροφική ασφάλεια και άλλοι τομείς. Επειδή είναι κοινή έκθεση, εδώ δεν εξετάζουμε μόνο το τι κάνουμε εμείς, αλλά δίνουμε έμφαση και στη συνεργασία, στις συνεργασίες επιτόπου στις χώρες αυτές, πώς τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συνεργάζονται επιτόπου στα πλαίσια της έντονας 2030, μια ατζέντα που έχουν συμφωνήσει τα κράτη-μέλη και αναπτυσσόμενες χώρες στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, Βεβαίω αυτό είναι σημαντικό και εν ώψη των διαπραγματεύσεων για, τα, για το επόμενο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, Όπω ξέρετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτείνει τον κοινό προγραμματισμό ω καλύτερο τρόπο συνεργασίας μεταξύ κρατομελών και Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Ορισμένε φορέ βέβαια δεν ακολουθούμε τον κοινό προγραμματισμό, ορισμένε φορέ έχουμε και κοινή εφαρμογή, κάποια προγράμματα εφαρμόζονται σωστά ε, ταυτόχρονα, από διάφορε εμπλεκόμενε φορέ και από την Ένωση και έχουμε και κάποια παραδείγματα εδώ και εκεί, στη Σενεγάλη, στην Κένια, κοινών πλαισίων αποτελεσμάτων. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη από κοινού φτάνουν σε μια συμφωνία με την χώρα εταίρο για το ποιο θα είναι το πλαίσιο των αποτελεσμάτων για το έγγραφο κοινού προγραμματισμού, παραδείγματο χάρη με την Κένια ή με τη Σενεγάλη. Επίσης προσπαθούμε να εργαστούμε πάνω σε νέα μέσα εξειδικευμένα όπως έχουμε πει και στην προηγούμενη συζήτηση για το σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων. Ε, Όμω σε επίπεδο αποτελεσμάτων είναι δύσκολο να δούμε ποιο είναι ο αντίκτυπο αυτών των νέων εξελίξεων. Πολλά από τα project τα οποία ξεκινάμε, για τα οποία ξεκινάμε να λαμβάνουμε κάποια αποτελέσματα, είναι project τα οποία είχαν προετοιμαστεί και είχε ξεκινήσει η εφαρμογή του πριν το 2015 ή εκεί κοντά Οπότε κατά κάποιο τρόπο είναι δύσκολο τώρα να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα τη επίπεδο SDG. Κάποια από τα SDG αυτά βέβαια είναι πολύ εστιασμένα και μπορεί κανεί να διαπορτήσει στον τομέα τη εκπαίδευση, παραδείγματο χάρη, αλλά είναι πολύ, πολύ πιο περίπλοκο όταν θέλουμε να περάσουμε σε ζητήματα όπω η ωκεανή, η βιομηχανοποίηση, οι ανισότητε κτλ. Τέλο, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή, την Επιτροπή σας, όχι μόνο για τη δυνατότητα που δίνετε σήμερα, αλλά για το γεγονό ότι έχετε δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα στην προώθηση τη Ατζέντα 2030, έχετε συνεργαστεί με τον Επιτροπή περιβάλλοντο. Αυτό δείχνει ότι πώ εφαρμόζει η Ένωση την Ατζέντα 2030 και βεβαίως ε, ε, αναμένουμε τη μονησία την έκθεση πρωτοβουλία, τη δική σα. και θα δούμε τι από αυτά μπορούμε εμείς να συμπεριλάβουμε ε, στις εργασίες μας κατά την ολοκλήρωση της κοινή ε, συγκεφαλαιοτικής έκθεσης. Ε, θα πρέπει βεβαίως να πάμε και στο φόρουμ ε, υψηλού επίπεδου τον Ιούλιο, θα γίνει και ένα άλλο φόρουμ το Σεπτέμβριο, είμαστε το 2019 είπαμε, είναι η χρονιά όπου ανεβαίνουμε επίπεδο, ε, μέσα και έχουμε την Υπουργική τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο είναι σύνοδος κορυφής πια, και γι' αυτό θα προχωρήσουμε, θα, θα προσπαθήσουμε κάποια αποτελέσματα της κοινή κεφαλική έκθεσης να τα παρουσιάσουμε εκεί με το έγγραφο διαβούλευση της Κομισιόν βέβαια. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια παρουσίαση όπου θα είμαστε θετικοί, επικοδομητικοί, θα δείξουμε τις δυνατότητε που έχουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστούν, αλλά και κάποιους τομείς όπου ε, θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση ή θα πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Είναι σημαντικό πάντως για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τον νέο Ευρωκοινοβούλιο να έχουν στα χέρια τους αυτή την κοινή κεφαλαιοτική έκθεση που είναι η πρώτη. Γι' αυτό το εξετάζουμε με τα κράτη-μέλη ε, για το πώς θα αντιδράσουν και αυτοί. Είμαστε όλοι στην ίδια κατάσταση, είμαστε δωρητές. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι ε, για τα SDG εμείς, ε, διότι τα προγράμματα αυτά σχεδιάστηκαν πριν τη θέση σε ισχύ ή κατά τη θέση σε ισχύ του 2030 δεν θα είναι όμω πια αυτό δικαιολογία το 2023 όταν θα κάνουμε τη δεύτερη εξυγκεφαλωτική έκθεση τότε δεν θα είναι απαράδεκτο η Κομισιόν, τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση να πούν και πάλι ότι δεν μπορούν να παρουσιάσουν κάτι συγκεκριμένο για τα SDG. Θα πρέπει λοιπόν να τα δούμε αυτά και να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ να απαντήσω σε ερωτήματα που ενδεχομένω να έχετε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ μαζί σας. Ευχαριστώ Λίντα. Να σας ενημερώσω κι εγώ με τη σειρά μου για το τι έχουμε ζητήσει εμείς ως Επιτροπή από τις αρχές του Κοινοβουλίου να κάνει για την παρακολούθηση των βιώσιμων στόχων. Συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, όπως ξέρετε. Την προηγούμενη εβδομάδα στη διάσκεψη των Προέδρων πήραμε την έκθεση και επειδή κάθε χρόνο οι πολιτικοί ρωτούν την Κομισιόν και τους υπουργού τι θα κάνουν για να μην χαθεί η όθηση και στην επόμενη θητεία θέλουμε που κάθε χρόνο να υπάρχει τον Ιούλιο ε, μια αντιπροσωπεία που θα την κυρίως από μέλη των Επιτροπών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αλλά και από άλλες επιτροπές ε, για το HRPF. Παραδείγματο χάρη τα θέματα των μεταφορών, η γεωργίας, αν τεθούν τέτοια θέματα, να έρχονται βουλευτές από αυτές τις επιτροπές, ώστε να καταλάβουν όλοι οι βουλευτές τι είναι οι στόχοι της ανάπτυξη, ανάπτυξης και με το κλίμα. Τι ετήσιες αυτές διασκέψει των συμβαλωμένων μερών, τα κόπα, που θέλουμε να κατατίθεται ψήφισμα από το Κοινοβούλιο. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση για να είναι υπόλογες οι διάφορες αρχές. Θα έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο των εργασιών των διαφόρων επιτροπών του Κοινοβουλίου για τους στόχους μίσης ανάπτυξης. Αλλά πρέπει πρώτα να το επικυρώσει η διάσκεψη των Προέδρων και μετά θα δούμε. Κυρίως οι βουλευτές που θα επανεκλεγούν εσείς που κατεβαίνετε στις ευρωεκλογέ πρέπει να μας βοηθήσετε. Για τη δελταντεύκο. Το βασικό είναι το πλαίσιο αυτή τη στιγμή, το πλαίσιο αναφοράς και κοινή συνεννόηση μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών για το πώς θα πρέπει να είναι αυτό το πλαίσιο. Ώστε μέχρι το 2023 τα μέτρα και η μέτρηση πρόοδου σε σχέση με τους στόχους του 2030 να είναι λίγο πιο απτά. Πότε θα έχετε την έκθεσή στον Απρίλιο, είπατε. Μέσα Απριλίου, μάλιστα. Τότε δεν θα συνεδριάζουν επιτροπές. Άρα να σημειώσουν ε, το προσωπικό να το σημειώσει για το επόμενο κοινό. Η Τζούντιθ. Καλό νέο. Έψαχνα τα χαρτιά μου. έλεγα κινήσει και οφαλωτική έκθεση. Μα δεν τη διάβασα. Α, δεν υπάρχει λοιπόν και γι' αυτό δεν την έχω διαβάσει. Ηρέμησα τώρα. Έχω όμως μια άλλη ερώτηση. Γιατί νομίζω ότι τα κράτη-μέλη της ε- Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε ό,τι αφορά τα συγκεφαλωτικά θέματα που έχουμε ένα πρόβλημα. Το Δεκέμβριο με την τελική ψηφοφορία στα Ηνωμένα Αθήνα, το Μαρακές. Είδα ότι οι Αυστριακοί απήχαν ευτυχώς, ενώ είχαν που θα καταψήφιζαν, αλλά αν κατάλαβα καλά και για άλλα θέματα, όπως αναπαραγωγικά δικαιώματα, σεξουαλικά δικαιώματα, πολιτικές που εμείς εδώ τις ψηφίζουμε ως ευρωπαϊκές, δεν στηρίζονται από κάποια κράτη-μέλη όταν ψηφίζουν στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Γι' αυτό έτσι κάπως εκμεταλλεύομαι αυτό το σημείο στη Μεσδιάταξη να θέσω αυτό το ερώτημα για να μου πείτε εσείς πώς μπορείτε να επηρεάσετε το κοινό προγραμματισμό και αυτή τη συγκεφαλαίωση. Πρόεδρος, κάποιος άλλος έχει να θέσει κάποιο ερώτημα σε αυτή τη φάση. Όχι, ο Φέλιξ τότε. Η Τζούντιθ βέβαια κάπως διεύρυνε το πλαίσιο και το φάσμα, αλλά σίγουρα το πολυμερές θεματολόγιο θέλουμε όλα τα κράτη-μέλη να το υποστηρίξουν, και απομακρυνόμαστε από άλλα τέτοια θεματολόγια που είχαν εγκριθεί το 2015 και στηρίζουμε αυτό που επίσης το 2015 εγκρίθηκε. Ο Φέληξ, ακούστε, σε ό,τι αφορά αυτή την κοινή συγκεφαλωτική έκθεση, το νόημα που έχει είναι να δει τι κάνουν τα κράτη-μέλη, τι κάνει η Ένωση και εμείς που εκπονούμε αυτή την έκθεση θα προσπαθήσουμε να είναι στο δυνατόν ευρύτερη κάτι μεταξύ περίληψης και αναλυτικής έκθεσης. Δεν είναι εύκολο, αλλά τέλος πάντων θα περιοριστούμε σε αυτά για τα οποία υπάρχει πλήρη συνένεση. Όπως είπατε και κάποια κράτη-μέλη δεν συμφώνησαν για το μεταναστευτικό ή για κάποια άλλα, όπως τα λένε οι ειδικές εκθέσεις, αλλά υπάρχουν άλλα κράτη που έχουν προωθήσει project σε αυτά τα θέματα. Και εκεί υπάρχουν δείκτες και στόχοι στο πλαίσιο του θεματολογίου του 2030, άρα δεν βλέπουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Να παρουσιάσουμε εμείς τι κάνουν από κοινού τα κράτη, αν είναι για την υγεία, αν είναι για την ε, ε, αναπαραγωγική υγεία, αν είναι για τις ισότητες, τέλος πάντων διάφοροι στόχοι, 4, 5, 10. Έτσι κάπως θα προχωρήσουμε. Και όσο περνάμε και στην επόμενη φάση, αλλάζουμε το στόχο. Το 2023 δηλαδή θέλουμε να είμαστε σε μια κατάσταση που να μπορούμε να κάνουμε πολύ πιο σαφείς αναφορές για τους δείκτες και τους στόχους και τους βιώσιμους ε, στόχους ανάπτυξης. Ε, αυτό δεν το βλέπετε τώρα. Υπάρχουν ομαδοποιήσεις κατά στόχο, αλλά όχι κατά βιώσιμο στόχο ανάπτυξης και δείκτη. Εμείς θα προσπαθήσουμε με τα κράτη-μέλη να συνεργαστούμε προς αυτό και αν περάσει και το NDCI θα έχουμε και τα κοινό πλαίσιο αναχώρα για να πούμε τοπικά τι γίνεται με τους βιώσιμους στόχους ανάπτυξης. Έχουμε ξεκινήσει επίπεδο για τη συζήτηση. Έχουμε το νέο development system και την ε, σχετική του μεταρρύθμιση και θέλουμε τη συνεργασία στο τοπικό επίπεδο να την ε, ενεργοποιήσουμε με γνώμονα το θεματολόγιο του 2030 για να μετρήσουμε τα αποτελέσματα. Αυτό είναι ο στόχο μα για το 2023. Αν δείτε τώρα τι κάνουν τα κράτη-μέλη εσωτερικά και εξωτερικά, έχουμε το σύστημα της ε, θελοντικής αναθεώρησης και έχουμε και το HLPF, το τέταρτο, ε, λίγη το Σεπτέμβριο, κλείνει τον πρώτο κύκλο, τον πρώτο τετραετή κύκλο από τότε που τέθηκε σε ισχύ το θεματολόγιο 2030 και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Και αν μπείτε στο Sustainable Knowledge Platform, στην ιστοσελίδα αυτή ε, του ΟΗΕ, θα δείτε αυτά τα voluntary annual reviews που έχουν καταθέσει τα κράτη-μέλη. 130 μέχρι στιγμής. Θα δείτε ότι σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη, 22 νομίζω, και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Και τα περισσότερα κράτη του 45 φέτος από τον μέχρι το Σεπτέμβρη θα έχει καλυφθεί το 90 95% των μελών ε, του ΟΗΕ που θα έχουν παρουσιάσει αυτές τις εκθέσεις. Αυτό είναι θετικό και πρέπει και εμείς να συγχρονιστούμε ως Ένωση και εσωτερικά και εξωτερικά. Και όταν ξεραστούμε το πρόγραμμα και την ψυχική συνεργασία θα το θέσω. Είναι μια Συζήτηση όμως που πρέπει να γίνει διαρθρωμένα. Και αυτός είναι ένα σημαντικό στόχος πολιτικός. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η Ρουμανική Προεδρία ξέρω ότι είναι πολύ δραστήρη. Του συζήτησα στην και υπάρχει κάποια ειδική επιτροπή και άλλες χώρες έχουν ειδικές επιτροπές. Καλό είναι πάντως τα μέλη της Επιτροπής μας να ξέρουν και τις εκθέσεις των δικών τους χωρών για να τις μελετήσουν. Ο Μισελ Γκέρενς θέλει κάτι να σας ρωτήσει. Έχω κι εγώ όμως μια ερώτηση. Για να είναι ορατό αυτό που κάνει ο θα πρέπει οι βουλευτές ε, από τις χώρες εταίρους επίσης να γνωρίζουν. Μάλλον δεν είναι όμως τόσο για το τι γίνεται στις χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νιγηρία, Κένια για παράδειγμα. Υπάρχουν ειδικέ επιτροπέ στα κοινοβουλιά του που μελετούν του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. Καλό είναι να βλέπουν και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα εθνικά σχέδια. Μισελ όμως, ήθελες κάτι να ρωτήσεις. Μία πολύ απλή ερώτηση σχετικά με τη μεθοδολογία. Ζητάτε λοιπόν συνεισφορές ε, από τις χώρες και εγώ θα ήθελα να ξέρω με ποια διαδικασία θα εγκριθεί η έκθεση. Φαντάζομαι ότι η συζήτηση θα γίνει σε αντιπαράθεση με τις χώρες μέλη και εάν ε, ε, ε, θέλετε εσείς να έχετε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, θα πρέπει και οι χώρες να έχουν κάποιο λόγο. Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα να πουν την άποψή τους. Αλλά θα ήθελα να με καθησυχάσετε όσον αφορά το εξή, ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν την άποψή τους. Η Κομισιόν έχει αρκετό κύρος έτσι ώστε να πει ότι αυτό είναι το σχήμα το οποίο θα αφορά και τους 28 και ε, με τον τρόπο αυτό να μην επιβληθεί ε, η άποψη ορισμένων κρατών μελών. Γιατί γνωρίζουμε ε, ότι συνήθως τα Υπουργεία θέλουν να παρουσιαστούν με το πιο καλακευτικό τρόπο. Αυτά. Ναι, είναι κάτι το οποίο θα ρωτήσουμε και στην έκθεσή μας. Δηλαδή ε, ότι η Κομισιόν δεν είναι μονάχα ένα γραμματοκιβώτιο στο οποίο ρίχνουν τις επιθυμίες τους και τα γράμματα που θέλουν να στείλουν τα κράτη-μέλη, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο και οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνεται σε τακτικά διαστήματα η αξιολόγηση της πρόοδου. Και, εν πάση περιπτώσει, εάν δεν το κάνουν τα ίδια θεσμικά, τα θεσμικά όργανα, θα το κάνουν άλλοι, π.χ. μη κυβερνητικέ οργανώσεις. και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα πρέπει ε, να λειτουργήσουμε ε, ως Ευρώπη στο σύνολο, συνολικά και όχι ως Γερμανία ή Γαλλία ή οτιδήποτε. Φέλιξ. Ευχαριστώ. Εμείς είμαστε ε, αρκετά τίμοι, έντιμοι σε σχέση με αυτά που ζητούν τα κράτη-μέλη και αυτό που μας ζητούν από μας τώρα βέβαια μπορεί να υπάρχει παράδειγμα μιας χώρας μέλους που παρουσιάζει κάτι ενδιαφέρον ή καινοτόμο, ας πούμε. Αυτό το μοιραζόμαστε με τα κράτη-μέλη. Αν το παράδειγμα δηλαδή είναι ένα παράδειγμα το οποίο εκείνοι οι ίδιοι, τα ίδια τα κράτη-μέλη θα ήθελαν ε, να πάρουν ως παράδειγμα και αν θέλουν να αλλάξουν την μεθοδολογία και το θεματολόγιο εργασίας τους. Αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο ε, στο οποίο εμείς αποφασίζουμε, δηλαδή εμείς αποφασίζουμε το παράδειγμα και όχι μόνο παραδείγματα τα οποία είναι καλά όσον αφορά το αποτέλεσμα, αλλά και παραδείγματα τα οποία είναι διδακτικά όσον αφορά την μεθοδολογία. Βεβαίως, οφείλω να σας πω ότι δεν έχουμε ακόμα αυτά αποτελέσματα και καμιά φορά, πώς να σας το πω, δεν έχουμε και αρκετή φιλοδοξία όσον αφορά τη μεθοδολογία, ας πούμε. Εγώ ε, σκέφτομαι να συναντηθώ με τα κράτη-μέλη ρωτώντας τους, ζητώντας τους να μου πούνε συγκεκριμένα πράγματα. Τι θα θέλατε να πουλήσετε στα, ε, ε, στα Ηνωμένα Έθνη τι θέλετε συγκεκριμένα να αλλάξετε στο θεματολόγιο του 2030, γιατί ε, δεν θέλουμε ε, να συνεχίσουμε με τα ίδια και τα ίδια. Να πάνε, θέλετε ας πούμε να συνεχίσουμε προγράμματα για τα κορίτσια που πρέπει να πηγαίνουν περισσότερο στο σχολείο ή θέλετε κάτι άλλο, θέλετε να αλλάξουμε την προσέγγιση, πείτε μου με ποιο τρόπο θέλετε να αλλάξουμε την προσέγγιση. Και για να απαντήσω στη Λίντα όσον αφορά τα κοινοβούλια. Εμείς επιμένουμε σε ένα σημείο ε, πολύ όσον αφορά αυτές τις εθελοντικές εθνικές επισκοπήσεις. Αυτές οι εκούσιες ε, αξιολογήσεις να γίνονται, να παρουσιάζονται ε, από τα κράτη-μέλη με την, με την μέγιστη δυνατή παρουσία εμπλεκομένων ενδιαφερομένων stakeholders θέματα τα οποία ας πούμε εμπλέκουν και πρέπει να εμπλέκουν και την κοινωνία θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται με την σχετική λογοδοσία ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών. Και έτσι ώστε να καθορίζονται και σωστά οι προτεραιότητες ε, υπό τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπου κυβερνήσεις ε, πήραν ε, μαζί τους ε, μεγα, πολυπληθή αντιπροσωπεία εμπλεκομένων βουλευτών, Εθνικού Κοινοβουλίου κλπ. Φανταστείτε ότι ε, το VNR, ε, στο VNR εκπροσωπούνται περίπου 120 ε, χώρες και φανταστείτε εκπροσώπους οι οποίοι, αντιπροσώπους μάλλον, οι οποίοι συνοδεύονται και από πολυπληθείς αντιπροσωπείες εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και επομένως αυτό κατά κάποιο τρόπο τους ε, επιβεβαιώνει και την ε, δύναμη που έχουν. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση του Γενικού Διευθυντού, να τον ευχαριστήσουμε για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε. Και άλλωστε θα τα ξαναπούμε όταν το Σεπτέμβρη η, αποστολή μας, ε, η Επιτροπή μας θα στείλει αποστολή στην Νέα Υόρκη. και οπωσδήποτε θα ζητήσουμε και βοήθεια, άλλωστε και τον Ιούλιο δεν θα είχε ξανασυσταθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις εκλογές. Προχωράμε πάντως και είναι πολύ ευχάριστο Okay, we're going to move on to item 7. I'm just asking the commission official to come. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Περιμένουμε τον ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι καλό να βλέπουμε μπροστά τους αυτόν που τους μιλάει στην ε, Επιτροπή μας, να μην μιλάει από πίσω. Δεν ξέρω αν θα έρθετε εδώ, θα μείνετε εκεί. Ωραία, περνάμε στο σημείο 7. Η κατάσταση στη δημοκρατία του Κονγκό. Μια χώρα για την οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές στην Επιτροπή μας και σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα δώσουμε Δώσαμε και το βραβείο Ζαχάροφ στον Δόκτωρ Μακουέγγι για το έργο του εκεί. Τώρα έχει και το Νόμπελ Ειρήνης. Είδαμε και τον Εμμανουέλ Ντεμερό, τον επικεφαλής του Εθνικού Πάρκου, για τη δουλειά που γίνεται εκεί. Δυστυχώ δεν μπόρεσα να είμαι εδώ. Έχασα εκείνη την παρουσίαση. Είναι πάντως ε, σημαντικά αυτά που συμβαίνουν εκεί. Και τώρα βεβαίως ε, το σημερινό θέμα είναι οι εκλογές στο Κονγκό που έγιναν ε, στην περίοδο των Χριστουγέννων. Οι συνάδελφοι θα γνωρίζουν ότι το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο. Από όσο ξέρω έχουμε προσωρινή ανακήρυξη αποτελεσμάτων, αλλά δεν είναι ακόμα σαφές το αποτέλεσμα θα αφήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση να τα εξηγήσουν και κάτι όμως που δεν ήξερα. Ο Μπαρτ Ούβε, ο πρέσβης της Ευρωπαϊκή Ένωσης ε, στο Κονγκό, του ζητήθηκε να φύγει στις 27 Δεκεμβρίου, από όσο ξέρω. Ενημερώστε, με, ενημερώστε μας ε, και από αυτού ποιο είναι το καθεστώ δηλαδή, τη αντιπροσωπεία μα εκεί αυτή τη στιγμή. Έχουμε δύο μιλητέ. Ο Χεράντο Χίλεν από την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, θα μα μιλήσει ενδεχομένω για τι εκλογέ και την παρακολούθησή του και η Φραντσέσκα Ντιμάρο θα μα πει για την ε, συνεργασία με την Δημοκρατία του Κονγκό σε αυτό το καθεστώ, σε αυτό το πλαίσιο πολιτικής αστάθειας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Χαίρομαι που βλέπω και κάποια γνώριμα πρόσωπα που συνάντησα και στις αποστολές ε, ε, στην Γουινέα. Χαίρομαι που, είναι εδώ, είμαι εδώ μαζί σας. Να πω δύο-τρία λόγια εισαγωγικά. Εδώ έχουμε βέβαια μια απλά, απλά ανταλλαγή απόψε, οπότε θα είμαι σύντομος. Να ξεκινήσω με τα δύο σημεία στα οποία αναφερθήκατε. Το συνταγματικό δικαστήριο κατόπιν προσφυγών. Τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακής ε, απέριψε αυτές τις προσφυγές και επίσης την ίδια, το ίδιο βράδυ, την ίδια νύχτα ανακοίνωσε το τελικό, το οριστικό αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Ο επικεφαλής ε, της αντιπροπίας μας ε, του ζητήθηκε τέλη Δεκεμβρίου να, να φύγει, να τον ανακαλέσουμε. Μας έδωσαν 48 ώρες για να το κάνουμε και του ζητήσαμε όντως να επιστρέψει στο, στις εγκαταστάσεις μας, στην έδρα μας. Θα δούμε τώρα πώς εξελιχθούν τα πράγματα. Ποιο ήταν ο λόγο για τον οποίο ζητήθηκε κάτι τέτοιο από, τις από τι αρχέ του Κονγκό. Είναι, αυτό έγινε μετά την απόφαση να επεκταθούν για άλλο ένα έτος ε, οι κυρώσεις. Τα περιοριστικά μέτρα ε, απέναντι σε κάποιους ε, πολίτες του Κονγκό. Μετά την παράταση λοιπόν αυτών των ε, κυρώσεων το Υπουργείο Εξωτερικών μας μίλησε για αντίμετρα και αυτό είναι το αντίμετρο στην προηγούμενη περίπτωση. Αυτό για τα συγκεκριμένα θέματα που θέσατε. Βεβαίως όπως ξέρετε ή μπορείτε να φανταστείτε παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις στο Κονγκό. Έγιναν εκλογές. Αυτό είναι θετικό από μόνο το ότι έγιναν εκλογές. δόθηκε δυνατότητα στον λαό του Κονγκό να εκφραστεί μέσω των εκλογών αυτών. Βεβαίως υπήρξαν δυσκολίες, υπήρξαν και ζητήματα έτσι τεχνικά, αλλά αυτό δεν επηρέασε τις ίδιες ε, τις εκλογές. Δηλαδή υπήρξε ε, μεγάλη συμμετοχή στις κάλπες, λαμβάνοντας υπόψη τις ε, ευρύτερες συνθήκες, ήταν αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Αυτό λέει και η ομάδα των παρατηρητών από την Αφρικανική Ένωση και την ΣΑΝΤΕΚ αλλά και από εθνικού παρατηρητές. Όμως ε, θα γνωρίζετε ίσως ότι έλεγα χώρα μια σύνοδος κορυφής ε, στις 27 στις 17 Ιανουαρίου στην Άντισα Μπέμπα με την ε, ομάδα αυτή του ΣΑΝΤΕΚ συμμετείχε και ο κύριος Καγκάμι από τη Ρουάντα, ο πρόεδρος δηλαδή ε, της Αφρικανικής Ένωσης για να συζητηθεί η κατάσταση στο Κονγκό αυτή η άτυπη σύνοδος ε, πήρε θέση στις 17 Ιανουαρίου όπου αμφισβητεί ανοιχτά την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και ζητεί ε, να σταματήσει η ε, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με δήλωσή του υποστήριξε αυτή την πρωτοβουλία. Έκτοτε όμως, όπως είπα, απαντώντας το ερώτημά σας, το Σάββατο το βράδυ, το Συνταγματικό Δικαστήριο πήρε την απόφαση να απορρίψει τις προσφυγές. Ο Φέλιξ Τσισικέντη λοιπόν ε, έχει πλέον ανακηρυχθεί πρόεδρος. Υπάρχουν επίσης κάποιες δυσκολίες ε, τεχνικές, αλλά η αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων ε, ακούστε έγινε δηλώσεις και από τις δύο αποστολές παρατηρητών και από διεθνείς ε, παρατηρητές ε, που αμφισβητούν τα αποτελέσματα αυτά. Μετά την απόφαση όμως του Σταγματικού Δικαστηρίου η Αφρικανική Ένωση αποφάσισε να αναβάλει την ε, αποστολή μιας αντιπροσωπείας ψηλού επίπεδου στην Κινσάσα. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Όπως θα αντιλαμβάνεστε, η, στην περιοχή αυτή ενδιαφέρονται πολύ ε, και βεβαίως ε, έχουμε πολλά προγράμματα ανάπτυξης εμείς εκεί προς όφελος των πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν τα αποτελέσματα των εκλογών να αποτυπώνουν τη βούληση των πολιτών. Εμείς είμαστε πάντα υπέρ της ειρηνικής ε, επίλυσης οποιασδήποτε διένεξης, οποιασδήποτε διαφορά, και πρέπει βεβαίως ε, να γίνει σεβαστό το δικαίωμα ε, της ειρηνικής ε, διαμαρτυρίας για όσου επιθυμούν να διαμαρτυρηθούν. Εμείς παραμένουμε ετέρη εταίροι της ε, Δημοκρατίας του Κονγκό. Δεν έχει σταματήσει σε καμία στιγμή αυτό. Η Φρανσίσκα Ντιμάρο, η συνάδελφο, θα αναφερθεί σχετικά. Επίση χρησιμοποιούμε την ευκαιρία αυτή το γεγονός δηλαδή ότι είναι, στη, είναι εδώ Αφρικάνοι Υπουργοί σήμερα και αύριο. Ξέρετε ότι λαμβάνει η χώρα ε, διάσκεψη υπουργική με την Ευρωπαϊκή Ένωση αύριο το πρωί. Στο περιθώριο λοιπόν αυτής της συνάντησης θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις με τους Αφρικανούς εταίρους μας πριν καθορίσουμε κάποια νέα θέση πριν να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Η Πατή εκπρόσωπος ε, συζήτησε το θέμα του Κονκό άλλωστε σήμερα το πρωί στην, ε, στο Συμβούλιο Εξωτερικών της Ένωσης. Αυτά μπορώ να σας πω εισαγωγικά και αναμένω την ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα θέσω σίγουρα Ερωτήσει. Οι συνάδελφοι από την Φρανσίκα από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξη. ε, φαντάζομαι ότι δεν θα έχετε πολλά να μα πείτε εφόσον δεν υπάρχει επίσημη απάντηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ευχαριστώ πολύ και καλό απόγευμα σε όλου. Ναι, έχουμε πολλά και μεγάλα προγράμματα, 620 εκατομμύρια περίπου ευρώ στο πλαίσιο του 11ου προγράμματο ανάπτυξη, επιπλέον Άλλε δημοσιονομικέ γραμμέ, ε, μια γραμμή τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. κτλ. Όλα αυτά αφορούν τη δημοκρατία του Κονγκό. Θα ήθελα να σα πω τι έχουμε κάνει, τι κάναμε εμεί για τι εκλογέ. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι θέσαμε στη διάθεση κάποια χρήματα, 20 εκατομμύρια, για την προπαρασκευή της εκλογικής διαδικασίας ε, προς τις αρχές, να τους πούμε ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα, εφόσον τα επιθυμείτε, τελικά δεν χρησιμοποιήθηκαν εξωτερικά, ε, εξωτερική χρηματοδότηση από πουθενά ε, και την ε, ε υποστήριξη της ΕΜΟΝΟΥΣΚΟ είπαν μπορούμε να τα κάνουμε, μόνιμα κάνουμε μόνοι μας τις εκλογές, δεν θέλουμε βοήθεια από εκεί πέρα δεν μπορούσαμε να στείλουμε εμείς ε, ομάδα παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό που προσπάθησαμε να κάνουμε είναι να υποστηρίξουμε τους παρατηρητές σε τοπικό επίπεδο 20.000 ε, ε, άμεσα, περίπου 40.000 έμεσα. Πρέπει να ξέρετε ότι το γεγονό ότι μπορούσαν να παρατηρούν αυτέ τι εκλογέ κάποιοι παρατηρητέ είναι ο λόγο ε, για τον οποίο δεν μπορούσαμε να έχουμε αυτή τη σκληρή θέση και να πούμε ότι ότι θα εκλεγεί σίγουρα ο, ο πρόεδρος ο υποψήφιος, ο πρόεδρος. Ε, ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη συμμετοχή των παρατηρητών. Ε, υπάρχει και μια πίεση έτσι εκ μέρους των πολιτών εμέσως. Βεβαίως ε, κάναμε πολλά, ε, πολλά προγράμματα εκπαίδευσης για τη συμμετοχή, αύξηση της συμμετοχής των γυναικών. Στο 7% τελικά η συμμετοχή δεν είναι τόσο άσχημα. Τώρα πέρα από τις εκλογές ε, εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμευόμαστε ε, να συνεργαζόμαστε για σημαντικά προγράμματα με μεγάλο αντίκτυπο. Αναφερθήκατε στην υποστήριξη στην Ανατολική, ε, Ανατολικό Κονγκό ε, με την Βιρούγκα. Είναι σημαντικό αυτό και για λόγους σταθεροποίησης να δώσουμε οικονομικές δυνατότητες για τους ανθρώπους που ζουν εκεί κοντά στα πάρκα, τα μεγάλα εθνικά πάρκα. Επίσης υπήρξε μαζική υποστήριξη για τι βασικέ υπηρεσίε στον τομέα τη υγεία, 175 εκατομμύρια στον τομέα τη υγεία, ε, πάνε κατευθείαν στην υποστήριξη ε, ανθρώπων για να έχουν πρόσβαση στι βασικέ ε, υπηρεσίε υγεία. Συνεχίζεται λοιπόν η συνεργασία μα και τα περισσότερα χρήματα έχουν ήδη δεσμευθεί, 85%. Ε, είμαστε προ το τέλο δηλαδή του προγράμματο. Τώρα θα πρέπει να δούμε, ανάλογα και με τα αποτελέσματα, είναι κάτι που θα συζητηθεί ε, η νέα κυβέρνηση που θα αναλάβει καθήκοντα, ε, ποια γραμμή θα ακολουθήσει, αν θα πάει προς μια ατζέντα μεταρρυθμίσεων, ε, εάν ε, μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε κάποιους τομείς όπως η αστυνομία, η δικαιοσύνη, ιδιαίτερα, ιδιαίτερα τομέα της δικαιοσύνης, εκεί σκοπεύαμε να προτείνουμε μεταρρυθμίσεις, τώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε, είναι κρίσιμη είναι κρίσιμο ωστόσο τομέας. Θα δούμε όμως βέβαια, θα εξαρτηθούν πολλά από τι είδου κυβέρνηση θα προκύψει και από την πολιτική μας αποτίμηση. Ναι, ο τομέας δικαιοσύνης ε, είναι πάντα σημαντικός. Ο κ. Μακουάγκη έλεγε πάντα ότι πρέπει να γνωρίζουν οι εγκληματίες ε, ότι τους περιμένει δικαιοσύνη ότι θα λογοδοτήσουν όταν έχουν βλάψει γυναίκες και παιδιά. Ε, δεν ξέρω αν κάποιο θέλει το λόγο, η Σεσίλ Κίνγκε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γιατί ήδη τα περισσότερα έχουν υποθεί. Αυτές οι εκλογές όμως αποτέλεσαν πολύ βαθιά πληγή για τον λαό του Κονγκό και είναι δύσκολο να μιλήσω γι' αυτό. Θα ήθελα να κάνω όμως κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη, οι κυρώσεις θα διατηρηθούν, αυτές οι στοχευμένες ε, κυρώσεις ε, απέναντι σε όσους ε, έχουν παραβιάσει ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και λόγω των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί στο Κονγκό. Θα διατηρηθούν λοιπόν αυτές οι κυρώσεις γιατί Ακόμα σήμερα ε, βλέπουμε ε, πολλούς από τους εγκληματίες αυτούς ε, να κυκλοφορούν αδιάφοροι. Δεύτερον, ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις εκλογές. Δηλαδή, υπάρχει κοινή θέση. Εάν ναι, ποια είναι αυτή η κοινή θέση. Αναφερθήκατε στο Συμβούλιο, το οποίο έλαβε χώρα σήμερα το πρωί, με τη Φεντερίκα Μογκερίνη. Μπορείτε να μας πείτε την έκβαση δηλαδή τι υπόθηκε σχετικά με την ε, λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Δημοκρατική, συγγνώμη, λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, ναι. Μαρία Χόιμπουχ. Ναι, ευχαριστώ. Αυτό που θα με ενδιαφέρει να μάθω είναι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από την αρχή είχε υπολογίσει ότι ενδεχομένως να υπήρχε νοθεία των εκλογών χειραγωγής του αποτελέσματος και που ε, τι κατάλαβε η ε, αποστολή, η ομάδα αυτή ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Αφρικανική Ένωση πώς κρίνει το αποτέλεσμα και τι μπορεί να κάνει. Θα ήταν πραγματικά να, πολύ έτσι, συναρπαστικό και ενδιαφέρον να ξέρουμε ποια είναι εκτίμηση για τις Αφρικανικές Ένωσες. Ευχαριστώ. Ποιος θέλει να απαντήσει. Α, Σεσίλα, αν μπορείς, σβήσε το μικρόφωνο σου. Σε παρακαλώ. Ε, παρακαλώ. Η ΑΕΔ καταρχάς. Ναι, ευχαριστώ. Η βασική έκβαση της φορεινής αυτής συνεδρίασης, ε, με βάση την μέρος που έλαβα, ήταν ότι πραγματικά επειδή υπάρχει αύριο η υπουργική διάσκεψη με τους Αφρικανούς ομολόγους, αξιοποιήθηκε αυτή η δυνατότητα ώστε στο περιθώριο να συζητηθούν οι αντιδράσεις και έπειτα θα διαμορφωθεί η κοινή θέση σε ό,τι αφορά τις τελευταίες εξελίξεις. Εμείς ήμασταν σταθεροί και συνεπείς και λαμβάνουμε υπόψη τις θέσεις και της ΑΝΤΕ και της Αφρικανικής Ένωσης και της περιοχής των μεγάλων λιμνών. Πάντοτε λοιπόν προσπαθούμε να τους ακούμε και να υποστηρίζουμε τις δικές τους δηλώσεις και διακηρύξεις. Άρα θεωρούμε ότι και στην προηγούμενη περίπτωση οι δηλώσεις αυτές ήταν προς σωστή κατεύθυνση, αντιλαμβάνονται σωστά δηλαδή το τι έγινε στο Κόγκο. Έξω και στηρίζουμε το τι είπε η Αφρικανική Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη. Το είπα και στην αρχή της πρώτης μου παρέμβασης, ότι και οι αποστολές παρατήρησης, ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εγχώρια ομάδα είχε πολύ σαφή άποψη για το τι έγινε. Εκεί βασίσαμε και τη δική μας ανάλυση των αποτελεσμάτων. Αν δείτε τις διάφορες εκθέσεις, φαίνεται να υπάρχει μία αντίφαση μεταξύ του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών και των αποτελεσμάτων των ε, περιφερειακών και βουλευτικών εκλογών. Δεν έχει τελειώσει η διαδικασία, παρότι το Σταγματικό Δικαστήριο τη νύχτα Σαββάτου προς Κυριακή ξέσουν τη μηγορία του. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις περιφερειακές και βουλευτικές εκλογές. Γιατί θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα του συσχετισμού δυνάμεων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Όπως βέβαια και το σχηματισμό της κυβέρνησης. Δεν θέλω να πρόβω σε κάποιες εικασίες. Αυτό που εμείς έχουμε ζητήσει είναι να υπάρχει διαβα... διαφάνεια προς τα αποτελέσματα και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων από τα εκλογικά τμήματα. και τα κέντρα συγκέντρωση των αποτελεσμάτων, ώστε να έχουμε την μέγιστη δυνατή διαφάνεια για να υπάρχει και η μεγαλύτερη δυνατή νομιμοποίηση για όσους εκλεγούν. Είναι ενδιαφέρουσες νομίζω οι εξελίξεις. από πλευρά Αφρικανική Ένωση ήταν πολύ έντονε οι απόψει και οι τοποθετήσει. Η απόφαση που ελήφθη δεν έχει οδηγήσει ακόμα σε αποστολή ψηλού επίπεδου. Υπάρχουν όμως ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Γίνεται η συζήτηση σε επίπεδο Αφρικανικής Ένωση τώρα και υπάρχουν ε, διαφορετικές απόψεις από τα, ε, πίσω από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή παρόμοια είναι η κατάσταση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμεί πρέπει να βρούμε μια κοινή θέση. Ιδίω για τα πολιτικά ζητήματα. Γι' αυτό και πρέπει να είμαι κάπως προσεκτικός σε ό,τι αφορά την ε, θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη σε σχέση με τη γραμμή που θα ακολουθήσουμε για το επόμενο υπόλοιπο της διαδικασίας σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. πρώτη ερώτηση το είπα. Παρατάθηκαν για ένα ακόμα έτος. Όταν μιλάμε για περιοριστικά μέτρα σε βάρο ιδιωτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη ανα πάσα στιγμή μπορούν να αναθεωρούν τέτοιε αποφάσει. Άρα υπάρχει και εδώ αυτή η δυνατότητα. Απλά είναι κάπω νωρί ε, για να συζητήσουμε τώρα τι θα συμβεί όταν θα έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Μπορούμε να το επαναξιολογήσουμε το θέμα όταν θα έχει, επαναλαμβάνω, λήξει η διαδικασία. Η απόφαση για τις κυρώσεις, σας πενθυμίζω, statement of purpose, δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς στα αγγλικά, δηλαδή ποιοι είναι οι λόγοι ε, που οδήγησαν στο να ε, επιβληθούν κυρώσεις σε συγκεκριμένους ιδιώτες. Είχε να κάνει με την ε, καταστρατής ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και του εκλογικού νόμου. Όλα αυτά θα αξιολογηθούν δεόντως μετά την, το πέρας της διαδικασίας. Απλά είναι πολύ νωρίς προς το παρόν. Ωραία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον, επομένως δεν υπάρχει επίσημη θέση από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δεν, έχει ολοκληρωθεί, λοιπόν, ε, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Θα παρακολουθούμε από κοντά το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ και που μοιραστήκατε μαζί μας αυτές τις θέσεις. Περνάμε στο σημείο 8, παραμένουμε στην Αφρική, θα συζητήσουμε για την Ερυθρέα. Δεν ξέρω αν θέλει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν να έρθει εδώ να μα τα πει επισήμω, Να εξηγήσουμε λίγο στου συναδέλφου ε, γιατί βάλαμε το θέμα αυτό στη μερίσια διάταξη, το θέμα αυτό για την Ερυθρέα. Συζητήσαμε ε, το θέμα της Ερυθρέας ε, και άλλες φορές και γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι η συνεργασία με την Ερυθρέα πάγωσε πριν από 12 μήνες, τότε που η Κομισιόν άρχισε να δίνει κάποια νέα στοιχεία συνεργασίας με την Ερυθρέα. Και τώρα προτείνει η Κομισιόν ε, μεγάλη στροφή στρατηγικής όσον αφορά τη χώρα αυτή. Σας ε, έχει δοθεί και κάποια ενημέρωση μέσω ε, σημειώματος από την Γραμματεία Παρακαλώ πολύ να εγκαταλείψετε ησύχω την αίθουσα. Έχετε χώρο έξω, άπλετο, που μπορείτε να συζητήσετε όσο θέλετε. Λοιπόν, αυτό που άλλαξε τους τελευταίους μήνες είναι ότι ε, υπήρξε αποστασιοποίηση μεταξύ... Ε, ε, προσέγγιση μεταξύ Ερυθρέας και Αιθιοπίας. of relations and the process of from the cold. Και επομένως ε, έχουμε ένα ξεπάγωμα των σχέσεων και έναρξη νέων διαδικασιών. Θα θυμάστε ότι είχαμε και ένα ενδεικτικό πρόγραμμα με αντίστοιχη χρηματοδότηση για την ε, Ερυθρέα Όμω, το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα δεν ε, ε, ολοκληρώθηκε, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Τώρα η Κομισιόν ε, μας λέει ότι αναλαμβάνει πλέον δράση για τη διερήνευση στην περιοχή και μέσω της μεταφοράς 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα στο Ταμείο για την Αφρική. Θα ακούσουμε λοιπόν πιο συγκεκριμένα θέματα και ε, με ποιο τρόπο κυρίως ε, δόθηκαν νέες δυνατότητες στους λιμένες. Επίσης, να μην ξεχνάτε, συνάδελφοι, ότι δεν είμαστε ακόμα απόλυτα σίγουροι για τις προϋποθέσεις ε, οι οποίες διέπουν την απελευθέρωση αυτών των πόρων. και επίσης ε, δεν ξέρουμε κατά πόσον οι εθνικές υπηρεσίες ε, έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν, να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια, ε, σε ποιο σημείο βρίσκονται τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Θα περιμένουμε λοιπόν να μας πούν οι εμπειρογνώμονες πρώτα την άποψή τους και μετά θα και εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε ερωτήσεις. υπεύθυνο για τις σχέσεις τη Ευρωπαϊκής Ένωση με τις χώρες της Δυτική Αφρικής. Και θα έχουμε και έναν εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ πολύ Λίντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε σήμερα εδώ. Ξέρετε ε, πόσο ε, προσφυλή μας είναι τα θέματα αυτά και πόσο θέλουμε να τα προχωρήσουμε. Ε, έγιναν όντως κάποιες σημαντικές αλλαγές ε, στην Ερυθρέα τους τελευταίους μήνες. Κυρίως η κοινή δήλωση φιλίας και ειρήνης τον Ιούλιο του 2018 μεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθρέας που κλείνει κατά κάποιο τρόπο μια πολυετή σύγκρουση. Ξέρετε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας επίσης τον προηγούμενο Νοέμβρη ήρε ε, το εμπάργο όπλων. Και επίσης η Ερυθρέα θα προεδρεύσει την, της διαδικασίας ε, ε, του Χαρτούμ, καθώς επίσης και το Φόρουμ Συνεργασίας Σομαλίας, Αιθιοπίας και Ερυθρέας η Ερυθρέα και ε, η Αιθιοπία πλέον ε, μπορούν να συνεργάζονται, έχουν ανοίξει ε, οι δρόμοι, έχουν ξαναρχίσει οι επικοινωνίες και έχουμε ελεύθερη προώθηση προϊόντων μεταξύ των δύο χωρών. Και οι δύο κυβερνήσεις, και αυτό έχει υπογραμμιστεί πολύ, ιδιαίτερα από την ε, κυβέρνηση της Αιθιοπίας, ε, είναι, έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν στην οδό της ειρήνης ε, και την σύσφυξη των εμπορικών και άλλων σχέσεων. Ε, όσον αφορά τον υψηλό διάλογο, θα σας τα πει ο Πάτρικ, αλλά εν πάση περιπτώσει οι δύο κυβερνήσεις ε, σκοπεύουν να πάρουν, ε, να κάνουν μεταρρυθμίσεις και να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση ανεργία και άλλων σοβαρών θεμάτων. Προς δεν έχουμε δει όμως κάποιες μεταρρυθμίσεις όμως έχει υπογραμμίσει η κυβέρνηση ε, την ανάγκη να δημιουργηθούν ε, οι προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες έτσι ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις. Εμείς προτείνουμε τώρα μία νέα προσέγγιση όσον αφορά την ε, Ερυθρέα. Αυτό ε, συζητήθηκε από την ομάδα εργασίας ε, της Αφρικής ε, του Συμβουλίου τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Πολιτική συνεργασία, λοιπόν, πολιτικός διάλογος με εθνικές υπηρεσίες, με ομάδες ανθρωπίνων οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά βεβαίως και συνεργασία όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση. Εδώ μιλάμε για ένα νέο σημείο εκκίνησης ε, και ε, προχωράμε βάσει των λεγόμενων αρχών εμπλοκής, principles of engagement, ε, πριν φτάσουμε στην πραγματική συνεργασία. Ε, και πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν δόθηκαν ε, ε, κονδύλια και αυτό ήταν ιδιαίτερο επιζήμιο για τον λαό της Ερυθρέας. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αν δεν άλλαζε θέση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έμενε πραγματικά στο περιθώριο όσον αφορά την χώρα Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ε, να ε, υπάρχει ε, η μέγιστη δυνατή εμπλοκή στην χώρα αυτή έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει αποτελέσματα. Είναι μια διαδικασία η οποία βρίσκει σύμφωνη και την Ερυθρέα. Βεβαίως κάθε μορφή συνεργασία θα πρέπει να προωθηθεί με ταχύτητα γιατί διαφορετικά ε, θα έχουμε τα κλασικά προγράμματα EDF και τις κλασικές ε, διαδικασίες, οι οποίες όμως από μόνες τους δεν θα μπορέσουν ε, να προχωρήσουν. Γι' αυτό προτείνει η Κομισιόν να μεταφερθούν 80 εκατομμύρια από την, από το ενδεικτικό εθνικό πρόγραμμα στο καταπίστευμα και βεβαίως είναι θέμα το οποίο θα συζητηθεί και στο Κοινοβούλιο. Αυτό θα σήμαινε ότι θα μπορούσαμε να παρέμβουμε σε τέσσερις τομείς. Πρώτον, στις υποδομές, δρόμοι κλπ. Δεύτερον, δημιουργία, θέση, δημιουργία θέσεων εργασίας, ε, κατάρτιση κλπ. Τρίτον, ε, οικονομικές μεταρρυθμίσεις σε συνεργασία και με το Διεθνές Ταμείο. Και τέλος, αναγνώριση της ε, σημασίας που ε, δίνεται και από τον λαό και από την ηγεσία της ε, χώρας ε, στην κοινωνική και λοιπή ενσωμάτωση και στο θέμα του, της πολιτιστικής συμπερίληψης. Σε λίγο θα συνεδριάσει η Επιτροπή για το καταπίστευμα και μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα πρόγραμμα 20 εκατομμυρίων που αφορά αποκατάσταση οδικού δικτύου. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, δηλαδή η διαδικασία λήψης απόφασης έχει ξεκινήσει. Και ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλη του μήνα θα επιβεβαιωθεί. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η καλύτερη οδός, όχι μονάχα για την Ερυθρέα και για άλλες χώρες και εξάλλου ταυτίζεται και ανταποκρίνεται στους στόχους του καταπιστεύματος. Αυτά που κάνουμε δηλαδή στην Ερυθρέα ανταποκρίνονται στους στόχους του καταπιστεύματος. Τέλος, ε, ο Επίτροπος ε, υπολογίζει αρχές Φεβρουαρίου να βρίσκεται στην Ασμάρα δεν έχει επιβεβαιωθεί ε, η ημερομηνία της επίσκεψης, αλλά οπωσδήποτε ε, μετά από την επίσκεψη ε, ευχαρίστως να ξαναέρθω και να σας ενημερώσω για την έκβαση αυτής της αποστολής επιτόπου. Και βεβαίω να επαναλάβω ότι πάντοτε είμαστε απολύτως δεσμευμένοι στη σωστή σας πληροφόρηση και ενημέρωση. Να ακούσουμε τώρα τον κύριο Σιμονέ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα απαντήσω σα όσα είπε ο Χάνς Στάουμπολ, γιατί τα εξήγησε πολύ καλά. Βλέπουμε, βιώνουμε πολλές αλλαγές στην περιοχή αυτή. Ειρνευτική συμφωνία, ειρνευτική διαδικασία μεταξύ Ερυθρέας Αιθιοπίας, που ε, ξεκίνησε πέρυσι τον Ιούλιο, αλλά και η τριμερής διακήρυξη και συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Αιθιοπίας, Ερυθρέας, Σομαλίας. το όλο σύστημα των συμμαχιών, αν θέλετε, και των σχέσεων που αναπτύσσεται, βλέπω να αλλάζει στην περιοχή και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, λόγω των τεκτενόμενων μεταξύ Αιθιοπίας ε, και Ερυθρέας, αλλά και γιατί μπορεί δυνητικά να επεκταθεί σε όλη την περιοχή και με τις περιφερειακές οργανώσεις ε, έχουμε ιδιαίτερες ε, επαφές Όπω ξέρετε, έχουμε λοιπόν δυνατότητα να δράσουμε και να παράσχουμε υποστήριξη. Κάτι σημαντικό για εμάς είναι ότι ναι, πράγματι, όσα συμβαίνουν εκεί μπορεί να είναι καταλήτης ε, για πολύ μεγάλες αλλαγές. Αλλά δεν μπορούμε να διαβάσουμε την κρυστάλλινη σφαίρα, άρα ε, ελπίζουμε το καλύτερο. Ελπίζουμε αυτές οι νέες σχέσεις Αιθιοπίας-Ερυθρέας να ανοίξουν ε, νέους ορίζοντες και ευκαιρίες στην Ερυθρέα που προχωρήσει σε εκθετικές ε, μεταρρυθμίσεις. Ε, οικονομικά ελπίζουμε και πολιτικά να δούμε κάτι ανάλογο. Βέβαια, μέχρι στιγμής ε, μόνο εικασίες μπορεί να κάνει κανείς. Ελπίζουμε τη διαδικασία αυτή να μπορέσουμε να την πλαισιώσουμε, όπως και την επανέναρξη της συνεργασίας που είχε κάπως ανασταλεί. Και θέλουμε έναν πολιτικό διάλογο με περιεχόμενο. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την ηγεσία της Ερυθρέας. Από την Ασημάρα γυρίσαμε με την... Έδειξε ότι υπάρχει διάθεση για πολιτική εμπλοκή, για ό,τι υπάρχει του στόχους, στόχου, οικονομικέ πολιτικέ μεταρρυθμίσει, ανθρώπινα δικαιώματα, μετανάστευση, το να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα σχετικά θέματα. θα είναι και η χώρα που θα προεδρεύσει τις δικασίες του χαρτών, όπως και ο Χάνς. Αυτές οι νέες λοιπόν σχέσεις θα πρέπει να πατάνε σε δύο πόδια. Το πρώτο, ότι ναι, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε και εμείς μια σημασία σε αυτή την προσέγγιση για να ε, υπάρξουν ε, εκ νέου ε, συγκοινωνίες, δρόμοι και τα λοιπά μεταξύ των δύο χωρών, αλλά τη δημιουργία συνεργασία επίσης και τον πολιτισμό θέλουμε να υποστηρίξουμε. Ένα αυτό και δεύτερον, πολιτικός διάλογος με περιεχόμενο όπως είπα και πριν. Είναι σημαντικό επίσης να δούμε σε τακτά διαστήματα κατά πόσο είναι μια έγκαιρη προσέγγιση αυτή. Και θα επανερχόμεθα στα κράτη-μέλη, σε εσά, για να βλέπουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Δεν είναι όμως μόνο ο πολιτικός διάλογος αυτό που θέλουμε, ξεκινώντας από την Ερυθρέα. Δεν είναι η μόνη πλατφόρμα συζήτησης, διαλόγου, για να έχουμε μια επαφή με την Ερυθρέα στα συστήματα που μας ενδιαφέρουν. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών θα γίνει μια αξιολόγηση σε ό,τι αφορά τη Οικουμενική Περιοδική Ανθεώρηση ε, στη Γενέβη για την Ερυθρέα, όπου να είναι ξεκινά αυτή η διαδικασία. Και εμεί μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ερυθρέα. Η κατάσταση ξεκολουθεί να είναι σχετική. Είναι μέλος, γίνεται μέλο και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Ερυθρέα. Οπότε θα του προτείνουμε να αναλάβουν ε, δράση. Έχουμε τη διαδικασία του Χαρτούμ που όπως γνωρίζετε είναι σημαντική για μας και την προηγούμενη εβδομάδα πήγε στην Ασμάρα μια αποστολή που προσπάθησαν να εξηγήσει του. Ε, ομολόγου μα εκεί τι διακυβεύεται με όλη αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να είμαστε έτσι κάπως ε, τολμηροί, αλλά θέλουμε να υπάρξει αυτή η ομαλή προσέγγιση αλλά ό,τι και αν κάνουμε δεν λησμονούμε και το μακροπρόθεσμό μας στόχο που είναι να στηρίξουμε τις οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα αυτή. Γιατί χρειάζεται αυτό το μετασχηματισμό. Με έντονη βέβαια στα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί η κατάσταση, όπως είπα, των ανθρώπινων δικαιωμάτων εμπνέει ακόμη μεγάλες ανησυχίες. Πρόεδρος, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος συνάδελφος το λόγο. Νόρμπερτ Νόιζερ και Τζούντιθ Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ και εγώ για τις ε, παρεμβάσεις για τις αναφορές αυτές. Πιστεύω ότι η αλλαγή στην Αιθιοπία πραγματικά είναι κάτι που κόβει την ανάσα. Και στην Αιθιοπία είχαμε δει ε, τα πράγματα με κριτικό μάτι και βλέπουμε ότι η κατάσταση τώρα πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να δραστηριοποιηθούμε τώρα τάχιστα στην Ερυθρέα για να δώσουμε στη χώρα αυτή μια ευκαιρία. Και σίγουρα με τον πολιτικό διάλογο θα πρέπει να εκμεταλλευτούν ε, την ευκαιρία και οι ίδιοι οι Ερυθρεανοί, γιατί θέλουν, ε, πρέπει να βελτιωθεί εκεί η κατάσταση. Αλλά και η Αιθιοπία πρέπει να βελτιωθεί, γιατί είναι ένα παράγοντα σταθεροποίηση, ο μεγαλύτερο παράγοντα σταθεροποίηση ε, και Νομίζω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε μια αναπτυξιακή πολιτική ε, σωστή ε, για την Ερυθρέα. Έχω μόνο μια ερώτηση σε ό,τι αφορά την πολιτική κατάσταση στην Ερυθρέα. Ε, σε ποιο βαθμό είναι αισθητή η βελτίωση. Και σε ό,τι αφορά τον αριθμό των μεταναστών ε, από τη μεθόριο ε, μεταξύ Ερυθρέας και Αιθιοπίας. Ε, τι μας αφήνει, τι ελπίδα μας αφήνουν τα νούμερα. Τι στοιχεία έχουμε. Κύριε Σαζεντίνη. Συζητούμε το θέμα της αναπτυξιακής βοήθειας και συνεργασίας με την Ερυθρέα και στο παρελθόν. Και θυμάμαι η Επιτροπή αυτή να λέει όταν το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα υπογράφηκε ότι δεν ήμασταν ικανοποιημένοι, θεωρούσαμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν τονιζόταν αρκετά ως όρος. Στη συνέχεια ε, το Συμβούλιο, η Επιτροπή EDF αγνόησε παντελώς τις ανησυχίες του και τις επιφυλάξεις του Κοινοβουλίου και δεν το κάνουμε συχνά, δεν εξάζουμε συχνά επιφυλάξεις για, για δαπάνες EDF ήταν μια αρκετά εξαιρετική περίπτωση. Τώρα, επίσης δυσκολευόμαστε με το Africa Trust Fund και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ελέγχει αυτή τη χρηματοδότηση. Και εδώ έρχονται μαζί αυτά τα δύο. Βεβαίως, τα 200 εκατομμύρια ευρώ στο Εθνικό Αντικτικό Πρόγραμμα για την Ερυθρέα ήταν δύσκολο να δαπανηθούν. Το γνωρίζαμε αυτό. και στο προηγούμενο EDF στο 10ο πάλι ήταν δύσκολο να δαπανηθούν διότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες όταν υπάρχει ένα σχέδιο υποδομή, ένα project και δεν είμαστε βέβαιοι ότι οι άνθρωποι ε, αυτοί ε, θα χρησιμοποιηθούν, που θα χρησιμοποιηθούν στο project θα χρησιμοποιηθούν από το στρατό, ε, δεν πρόκειται να, δαπανίσουμε. Οπότε δεν θα πανούσαμε πολλά στο 10, οπότε δεν θα πανούσαμε και στο 11. Όμως μας έλεγε η διασπορά της Ερυθρέας, τι συμβαίνει εδώ. 200 εκατομμύρια ευρώ για τον Ασμάρα ε, με αυτή τη συμπεριφορά. Δεν δαπανήθηκαν τα χρήματα λοιπόν. Και προτείνατε στο Συμβούλιο και βεβαίως εκεί το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ελέγξει αυτά τα 180 εκατομμύρια που περισσεύουν από το EDF να, πάει στο, να πάνε στο Africa Trust Fund, διότι είναι πιο εύκολο να δαπανηθούν. Α είμαστε όμω ειλικρινεί εδώ, έτσι. Όχι μόνο επειδή είναι πιο γρήγορο, είναι πιο γρήγορο, αλλά πραγματικά τι σημαίνει αυτό. Δεν ελέγχει πια ούτε το Κοινοβούλιο, ούτε το Συμβούλιο για να μπορέσετε να δαπανίσετε αυτή την αναπτυξιακή βοήθεια γρήγορα. Πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Δεν είδαμε όμω να συμβαίνει κάτι στην Ερυθρέα ακόμα. Σε ό,τι αφορά το στρατιωτική θητεία. Αυτό που συμβαίνει στην αιθιοπική πλευρά είναι πολύ καλά νέα, βεβαίω, Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι καλό για την περιοχή, αν θέλουμε να βοηθήσουμε την Αιθιοπία, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Όμως, το να δαπανίσουμε τα χρήματα αυτά, ξεχνώντα τις προϋποθέσεις, του όρου που έχουμε θέσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί δεν βλέπω πώ θα μπορέσουμε να το σεβαστούμε αυτό, αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Εάν το πρώτο project λοιπόν είναι το, το θέμα του δρόμου, βεβαίως ο δρόμος μεταξύ των δύο αυτών ε, χωρών είναι, είναι εξαιρετικά σημαντική συμβολική σημασία. Όταν χτίζουμε ένα δρόμο, πολύ συχνά χρησιμοποιείται αυτή, αυτό το εργατικό δυναμικό που είναι σκλάβη στην πραγματικότητα. Πώς θα γίνει λοιπόν να μην συμβεί αυτό. Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπος Ανάπτυξης είχε στείλει μια επιστολή στον Ασμάρα και τον ρωτούσε τι έγινε με τον Ντάβιτ Ίσακ και δεν λάβαμε από όσο ξέρω ούτε καν απάντηση που να λέει ότι λάβαμε το γράμμα σας. Από πού λοιπόν έρχεται αυτή η ιδέα ότι αυτό θα βοηθήσει το καθεστώς της Ερυθρέας να βελτιώσει την κατάσταση των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Και τώρα είμαι όλο και πιο κοινική βέβαια. Μήπω εξακολουθούν να είναι μέρο τη διαδικασία του Χαρτούμ και μήπω επειδή προεδρεύουν τη διαδικασία του Χαρτούμ που είναι τόσο σημαντική για μα για τα ζητήματα μετανάστευση, που είμαστε διατεθειμένοι να παραβλέψουμε κάποια ζητήματα. Ξέρω ότι είναι κοινικό αυτό που λέω, αλλά δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό σας. Βλέπω γρήγορες, γρήγορο ξόδεμα χρήματο, χρημάτων για ένα καθεστώς το οποίο είναι η Βόρεια Κορέα της Αφρικής. Έως τώρα λέγαμε δαπανούμε μόνο όταν σέβεστε ε, τα, τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα το ξεχνάμε και αυτό. Η, η κυβέρνηση της Ερυθρέας ενδιαφέρεται για τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι που έχει ενδιαφέρον δεν ενδιαφέρονται οι ίδιοι να πλουτίσουν. Τι, γιατί λοιπόν θα κάνει τη διαφορά αυτό και, και επισήμω ποια είναι η ανακοίνωση δική μας. Δεν βλέπω δηλαδή πώς, και τελικά πώς το μάθαμε εμείς και όλο αυτό. Ναι, σε ό,τι αφορά τη μεταφορά στο Trust Fund, ναι, είναι σημαντικό να καταλάβουμε τη διαδικασία θα περάσει στην Επιτροπή EDF, φαντάζομαι, για να ζητήσετε η χρηματοδότηση αυτή να, να περάσει στο Trust Fund. Και μετά βεβαίω να δούμε και τι γίνεται στο Trust Fund. Σε ποια φάση βρίσκεται, βρίσκεται αυτή η, η διαδικασία. Καταλαβαίνω αυτά που λέτε για το καθεστώς. Ε, κάποιοι θέλουν να είναι πιο ανοιχτοί, κάποιοι όχι θέλει να ξεκινήσει ένα διάλογο με αυτό το καθεστώς. Πώ όμως αυτές οι δαπάνε ε, θα χρησιμοποιηθούν και τι θα γίνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Εφόσον δεν αλλάζει κάτι στην Ερυθρέα, ε, θα ρωτάει ο κόσμο γιατί να δίνουμε χρήματα σε ένα καθεστώ όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σε τραγική κατάσταση και, ότι, και όπου υπάρχουν σκλάβοι. Δεν μπορούμε να δώσουμε όλα αυτά τα χρήματα με τη μία. Θα παρακολουθούμε λοιπόν αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω ποιο θέλει να απαντήσει πρώτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, ναι. ναι ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και για την συζήτηση αυτή που έχουμε. Για το πρώτο που είπατε, που είπε ο κύριος Νόισερ, τα τελευταία στοιχεία που έχουμε για τη μετανάστευση από την Ερυθρέα δείχνουν ότι από το Σεπτέμβριο πέρυσι, το Σεπτέμβριο του 2018 δηλαδή, που, υπεγράφηκε η Ειρηνευτική Συμφωνία και άνοιξαν τα σύνορα, είχαμε 20.000 αφήξεις στα βασικά κέντρα ε, υποδοχής. Τώρα μιλάμε όμως πλέον για 250 250 άτομα, 280 τη μέρα ε, που φεύγουν από την Ερθρέα. Είναι αρκετά σημαντικά τα στοιχεία. Τώρα, για το θέμα που έθεσε η Ιούντιτ. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι η θέση του Κοινοβουλίου ελήφθη υπόψη από τα κράτη-μέλη, διότι επέμειναν στην αρχή της δέσμευσης και εφόσον ε, ακολουθούμε την αρχή της δέσμευσης δεν μπορέσαμε να δαπανίσουμε ούτε ένα ευρώ. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή υπήρξε αναστολή και μη πληρωμή. Σημειώσαμε αυτό που είπατε. Έχει αναγνωριστεί πολλές φορές ε, σε πολλά φόρουμ ότι υπάρχει έλλειψη ε, παρακολούθηση από το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά το Trust Fund. Το Κοινοβούλιο έχει το ρόλο του παρατηρητή ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε βεβαίως όλες τις πληροφορίες που θέλετε για αυτά που προτείνουμε, προτιθέμεθα να κάνουμε. Πώ λαμβάνετε πληροφορίε τώρα για αυτά για αυτή την αλλαγή. Πώς το μάθατε. Εμείς τηλεφωνήσαμε στη Λίντε, ε, Λίντα πριν από δύο εβδομάδες, είπαμε ε, καλό να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Έχουμε έρθει εδώ εθελοντικά να συζητήσουμε μαζί σας και θέλουμε να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Για να είμαστε σαφείς. Πώς ε, αυτή η υποστήριξη θα δομηθεί. Έχουμε παράλληλη ε, διαδικασία. Συνεργασία για την ανάπτυξη και πολιτική διαδικασία. Αν σε έξι μήνες ε, ε, δούμε ότι ο Πάτρικ και οι συνάδελφοι βρίσκουν τείχο μπροστά του και δεν προχωράνε, δεν προχωράει το θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στη Γενέβη, αν δούμε ότι ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε δεν έχει κανένα αντίκτυπο σε ό,τι αφορά τη βούληση τη κυβέρνηση εκεί να μεταρρυθμίσει τα, του στρατιωτική θητεία, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η προσέγγιση. Εμείς προτείνουμε 20 εκατομμύρια για οδικά έργα. Θα πάμε στην Επιτροπή EDF το Μάρτιο. Θα ζητήσουμε αυτή τη μεταφορά. Ε, αυτό σημαίνει πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί πέρα Απρίλιο-Μάιο, εφόσον λάβουμε το πράσινο φω. Οπότε έχουμε εδώ χρόνο μπροστά μα για να αξιολογήσουμε τι συμβαίνει σε αυτό το χρονικό διάστημα. Πρέπει επίση να παραδεχτώ ότι εάν δεν προχωρήσουμε με την κυβέρνηση τη Ερυθρέα, Μπορούμε να κάνουμε άλλα πράγματα με τα χρήματα αυτά στο Trust Fund. Αυτό είναι το καλό με το Trust Fund. Εάν δηλαδή δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε ε, τα project αυτά, θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά ε, σε ένα άλλο πλαίσιο, στο... για τους πρόσφυγες παραδείγματος χάρη, ε, έχουμε δηλαδή μια κάποια ευελιξία με το Trust Fund. Δεν συζητήσαμε λεπτομερώς με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης πώς θα παρακολουθήσουμε αυτές τις δύο διαδικασίες και πώς θα δώσουμε αναφορά γι' αυτό. Πάντως θα συμβεί αυτό και όποτε θέλετε ερχόμαστε στην Επιτροπή αυτή να σας εξηγήσουμε τι κάνουμε, να σας ενημερώσουμε για το project του Trust Fund. Και τέλος, δεν είναι δίκαιο νομίζω να πείτε ότι το Συμβούλιο ε, ανησυχεί ε, για το Trust Fund. Είχα μια συζήτηση για ε, την έκθεση του Μετρικού Συνεδρίου στο Συμβούλιο την προηγούμενη φορά και πραγματικά ήταν πολύ θετικά τα κράτη-μέλη. Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ θετικά στο το Trust Fund. Σίγουρα δεν ανησυχούν πάντω για την έλλειψη διακυβέρνηση στο Trust Fund. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ό,τι κάνουμε στο Trust Fund είναι αποτέλεσμα μια συζήτηση στην Επιτροπή, ε, στην Διοικητική Επιτροπή όπου συμμετέχουν ε, τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Σταματάω εδώ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι με τι εξωτερική δράση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τι αλλάζει στην Ερυθρέα. Ε, όχι πολλά, είναι αλήθεια, από επίσημης πλευράς. Γίνονται συζητήσεις για μεταρρυθμίσεις, συζητήσεις για νέα σχέδια, για την ε, στρατιωτική θητεία. Τι αλλάζει όμως, ήμουν εκεί, ήμουν και στο βορρά, έτσι, στο βόρειο μέρος της χώρας. Βλέπουμε ότι ανοίξαν τα σύνορα. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους κάτοικους της Ερυθρέας να μετακινηθούν, να ταξιδέψουν, να περάσουν τα σύνορα και να δουν πώς είναι να ζει κανεί. Ε, σε υπό ένα καθεστώ κάπως πιο ανοιχτό, σε μια κάπω καλύτερη κατάσταση. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Όταν λέμε λοιπόν ότι θα βάλουμε χρήματα στην Ερυθρέα, θα ρίξουμε χρήματα στην Ερυθρέα, δεν είναι αυτό ακριβώ αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και διορθώστε με αν κάνω λάθο. Θέλουμε να βάλουμε χρήματα για την ε, επαναπροσέγγιση μεταξύ Αιθιοπία και Ερυθρέα. Και η... αυτό μα το ζητάνε οι Αιθίωπε. Ε, θέλουν να συμβεί αυτό δεν μας ζητούν να, να βάλουμε χρήματα στην Ερυθρέα διότι ε, είμαστε ρεαλιστές ε, και αυτοί είναι οι ρεαλιστές στην Αιθιοπία ε, δεν βλέπουν να συμβαίνουν αλλαγές σύντομα είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί πρέπει δηλαδή, να προσκύσουμε πολύ προσεκτικά το θέμα της Ερυθρέας διότι ως Αιθίωπες δεν έχουν κανένα συμφέρον να καταρρεύσει η χώρα ε, Θέλουμε λοιπόν εμείς να στοιχηματίσουμε, να ποντάρουμε αν θέλετε, στην προσέγγιση των δύο χωρών. Η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορία των προσώπων, όσων είναι ανοιχτά τα σύνορα τουλάχιστον, διότι υπάρχει και το σενάριο ότι βλέποντας την επικαιρνότητα για τη, βιώσιμα, για τη, βιωσιμότητα του καθεστώτος να κλείσουν τα σύνορα εκεί στην Ερθρέα Για την ώρα δεν συμβαίνει αυτό. Ακούμε λοιπόν τους Αιθίωπες, ε, ακούμε γενικότερα την περιοχή. Θέλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην προσέγγιση μας. Βεβαίω μπορεί να μην μα πιστέψετε με βάση τα καλά μας λόγια και τις υποσχέσεις μας. Ζητήστε μας να, να ξανάρθουμε όμως, να σας πούμε τι έχει γίνει ε, ενδιάμεσα. Ενδεχομένω να μην έχει αλλάξει τίποτα σε έξι μήνε. Και τότε θα πρέπει να πάρουμε κάποια άλλη απόφαση, να κάνουμε κάτι άλλο με τα χρήματα αυτά. Θεωρούμε πάντως πω είναι πολύ δύσκολο να μην κάνουμε κάτι τώρα διότι υπάρχει μια ειρηνευτική διαδικασία μετά από 20 χρόνια χωρίς πόλεμο ούτε ειρήνη ξεκινάει μια ειρηνευτική διαδικασία δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη εμείς και να πούμε μας δεν μας ενδιαφέρει το θέμα αυτό λοιπόν για τα 207 εκατομμύρια ε, θέλω να προσπαθήσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε να πιάσουν τόπο να δούμε αν μπορούν να υποστηρίξουν αυτήν την ειρηνευτική διαδικασία αυτό που με εξέπληξε ε, στην Ερυθρέα είναι ότι παρά τις κατηγορίες που μας απευθύνουν, ε, διότι ήμασταν σκληροί μαζί τους και τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλα αυτά, εξακολουθούν να έχουν συμφέρον και να ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί μας. Περισσότερο από ότι με τους Κινέζους ή με τις χώρες του κόλπου. Έτσι λένε τουλάχιστον. Πάντως ε, είμαστε ακόμα στην αρχή και θα επανέλθουμε σύντομα να σας πούμε ποιε είναι οι εξελίξει. Τζούλη, θε να προσθέσει κάτι. Ναι, δύο, δύο πράγματα. Ένα. Ε, δίνετε έγκαιρα αυτά τα εργαλεία και χαίρομαι που τα λέτε στο Κοινοβούλιο. Αλλά δεν θα μπορούσατε να κάνετε στο χαρτί γραπτά την ανάλυση που κάνετε για το Συμβούλιο. Αυτό θα μας βοηθούσε πολύ. Επίσης, ερώτηση στη Λίντα και την Γραμματεία. Εάν δούμε από το EDF να πηγαίνουν κονδύλια στο καταπίστευμα πέρα και άσχετα από την κατάσταση στην Ερυθρέα τι γίνεται, γιατί εμείς ε, κατά κάποιο τρόπο ελέγχουμε το EDF. Δώστε μας λοιπόν γραπτά τις πληροφορίες αυτές, γιατί διαφορετικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, κατανοήσουμε πλήρως και ε, τις τελευταίες ε, αποχρώσεις, ας πούμε, της, των όσων μας λέτε προφορικά. Επίσης, θα πρέπει να ζητηθεί κάποια συμφωνία μεταξύ της χώρας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αυτόν τον τρόπο, είτε γίνεται η δαπάνη είτε όχι, η χώρα ξέρει τι είναι ουσιαστικό. Και γιατί λοιπόν η Ερυθρέα δεν λέει μέχρι τώρα είμαστε καλοί μαθητές, συνεργάσιμοι και εμείς θέλουμε λοιπόν οι δαπάνες να γίνουν μέσα από το ενδεικτικό εθνικό πρόγραμμα. Γιατί λέτε εάν δεν μπορούν να δαπανηθούν μέσω του καταπιστεύματος, τότε το βγάζετε από την Ερυθρέα και τα χρησιμοποιείτε κάπου αλλού. Αλλά αυτό δεν είναι πολύ ελκυστικό για την Ερυθρέα, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη. Τι κρύβεται λοιπόν πίσω από αυτό, γιατί η Ερυθρέα λέει ναι, ε, μπορεί να αποφασίσει αν θέλει ή δεν θέλει. Και εάν δεν τους δίνει τη δυνατότητα να δαπανίσουν κονδύλια του EDF, πώς μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα δαπανηθούν τα όσα περιλαμβάνονται στο καταπίστευμα. Okay, the paper. Όσον αφορά τα έγγραφα. Ε, υπάρχει ένα background note. Ναι, ναι, εξαιρετικό, λέει η κυρία Σαργεντίνη ε, και ε, γράφτηκε από την γραμματεία, δεν είναι έτσι. Η γραμματεία έδωσε γραπτά κάποιες εξηγήσει, αλλά εγώ θα ήθελα να δω τη, τα, τα, βασικά στοιχεία επί των οποίων βασίζονται οι λήψεις αποφάσεων, κομισιόν προς συμβούλιο. Θα δούμε, λέει η Πρόεδρος εάν μπορεί να μοιραστεί ας πούμε μαζί μας κάποιες προϋποθέσεις ε, κλπ. Για το ρόλο του καταπιστεύματος είμαστε παρατηρητές. Δεν είμαι σίγουρη πότε θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση. Για απαντήστε υπό τον έλεγχο του θεσμικού μου φύλακα, ε, ναι, θα μπορούσαμε, θα μπορούσαμε να ε, συγγράψουμε έτσι ένα υπόμνημα όσον αφορά τα θέματα τα οποία αναφέρατε. Σχετικά με την ε, ownership, την οικειοποίηση και το καταπίστευμα, είναι γεγονός ότι το γεγονός που, ότι χρησιμοποιούμε ε, το καταπίστευμα με κανένα τρόπο δεν ε, δυναμητίζει την οικειοποίηση από πλευράς της Αιθιοπίας. Εμείς ε, δεν θα μπορούσαμε να υποβάλουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα στην Operating Committee εάν δεν είχαμε πάρει τα μέτρα μας πριν. Γιατί προτείνουμε να προχωρήσουμε. Ναι, γιατί υπάρχει ανάγκη ευελιξίας. Εάν ε, δεν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο μέσω του Εθνικού Ενδεικτικού Προγράμματος, τότε θα είμαστε υποχρεωμένοι να δαπανίσουμε 3, 4, 5 μήνες ε, προσπαθώντας να επιτύχουμε κάτι, λαμβάνοντας τα υπόψη ότι τα κράτη-μέλη δεν ε, προβληματίζονται ιδιαίτερα με τη χρήση του καταπιστεύματος και λαμβάνοντα υπόψη ότι η άλλη πλευρά κατανοεί και τα θέματα διακυβέρνηση και τα προβλήματα και αυτά, ε, πήραμε αυτή την απόφαση. Δεν νομίζω ότι δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Εάν θέλουμε να ε, κινηθούμε έγκαιρα και σωστά, δεν αρκεί το EDF. Δεν είναι το, το, καλό, το καλύτερο δυνατό εργαλείο του EDF. Και επίσης να σας πω ότι έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί η άλλη πλευρά δεν δέχεται ε, ε, ή δέχεται με μεγάλη δυσκολία τις ε, στάνταρ διαδικασίες και μεθοδολογίες εργασίας που έχουμε. Τώρα, εσείς ίσως, και μια και είδαμε ότι δημιουργείται έτσι ένα άνοιγμα, γιατί δεν πάει το κοινοβούλιο επιτόπου να μιλήσει μαζί τους. Νομίζω ότι πραγματικά θα μπορούσαμε να σας υποστηρίξουμε και να βρούμε έναν τρόπο ε, αναφοράς ε, σε τακτά διαστήματα. Ναι, τι να σας πω τώρα, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να πάει κανείς να οργανώσει αποστολή εκεί. Τώρα έχουμε ε, το ζήτημα του νέου κοινοβουλίου κτλ. Κάποιοι συνάδελφοι είχαν πει ότι ήθελαν να, να οργανώσουν αποστολή στην Ερυθρέα, αλλά μας απέτρεψαν. Ωραία, άλλες ερωτήσεις, κύριε Σαργεντίνη. Μια πρόταση. Ε, ούτως ή άλλως ε, δεν υπάρχει χρόνος πλέον σε αυτή τη θητεία, αλλά ε, το να πάει μια αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου με ιδιαίτερη πολιτική κατάσταση ε, ε, ε, μια τέτοια επίσκεψη είναι πολύ ευαίσθητη εάν δεν έχουν υπάρξει προηγουμένως κάποια, κάποια μηνύματα αλλαγής από την άλλη πλευρά γιατί διαφορετικά θα είναι σαν να επικυρώνει κανείς τα όσα συμβαίνουν στη χώρα αυτή. Πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει την επόμενη Επιτροπή Ανάπτυξης και τους επόμενους συντονιστές. Θα δούμε ποια θα είναι τα μέλη της Επιτροπής τον επόμενο Ιούλιο. Ωραία, αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε και είναι πάρα πολύ θετικό που μας ενημερώσατε και ενημερώθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, τελευταίο σημείο για σήμερα το 8, που δεν ε, πιστεύω θα μας πάρει πολύ χρόνο. Είναι ουσιαστικά ομάδα παρακολούθηση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μετά τη Συμφωνία του Κοτονού. Ενημέρωση λοιπόν για την ε, συνεδρίαση που έγινε πριν από δύο εβδομάδες στις Βρυξέλλες. Είναι μια νέα ομάδα αυτή όπως γνωρίζετε η συμφωνία του Κοτονού λήγει το Φεβρουάριο του 2020, οπότε τώρα διαπραγματευόμαστε τη διάδοχο συμφωνία. Θέλουμε να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσει αυτές ε, και να τις παρακολουθεί. Εξού και δημιουργήθηκε μια ειδική ομάδα με μέλη από τις Επιτροπές ΑΦΕΤΙΝΤΑ, ΝΤΕΒΕ φυσικά και την αντιπροσωπεία στην Σωμή Κοινοβουλευτική Συνέλευση και Ευρωπαϊκή Ένωση και την αντιπροσωπεία στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα αναπτυξιακά θέματα. Έχουμε λοιπόν αυτή την ειδική επιτροπή παρακολούθησης, ε, γιατί όποιο και αν είναι το τέλο αυτής της διαδικασίας, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του, ε, τη σύμφωνη γνώμη του, οποιαδήποτε διάδοχο συμφωνία, τη συμφωνή Τελικά ήταν στο Στρασβούργο. Όχι την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν την Τρίτη, την προηγούμενη. Είχε έρθει και ο Επίτροπο ε, Μίμητσα να μιλήσει. Είναι ο επικεφαλή τη διαπραγματευτική ομάδα. Ε, ήταν μια ανταλλαγή απόψεων και κλεισμένων των θυρών για το τι συμβαίνει. Ήταν γενικόλογα αυτά, για να είμαι ειλικρινή, που ακούσαμε. Δηλαδή, ακούσαμε ότι υπάρχει συμφωνία τώρα μεταξύ ΑΚΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε ό,τι αφορά τη δομή και στρατικές στρατηγικές προτεραιότητες ε, το σκέλος ΑΚΕ δέχτηκε μια δομή με πυλώνες, να υπάρχει δηλαδή ένα, μια κοινή βάση και τρεις περιφερειακοί πυλώνες. Θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τους περιφερειακούς πυλώνες το Φεβρουάριο με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί το καλοκαίρι. Εμείς ε, όμως ε, δεν θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τα τεκτενόμενα, δεν θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από τις εκλογές και θα πρέπει να προετοιμάσουμε το έδαφος για το επόμενο κοινοβούλιο, τον Ιούλιο. Συνεχίζονται λοιπόν οι συζητήσεις. Από ό,τι γνωρίζουμε και στην Αφρική γίνεται μια συζήτηση για το κατά πόσο θα είναι μια Παναφρικανική Συμφωνία με Αφρικανική Ένωση και Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θα είναι ε, με την Υποσαχάρη Αφρική κτλ. Είναι η Μαρία, όχι, ο Νόρμπερτ ε, ήταν ο εισηγητή μα για τη μετά το Κοτονού. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι ή να, να δώσω το λόγο στη Μαρία να θέσει την ερώτησή τη Πρώτα η Μαρία ή η Νόρμπερτ. Ε, ο Νόρμπερτ Νόιζερ. Δεν υπάρχουν και πολλά που μπορώ να προσθέσω γιατί ήταν σιγαστικά σαφή αόριστα αυτά τα οποία συζητήσαμε την προηγούμενη πέμπτη λέει τώρα. Εγώ δεν ήμουν καθόλου ικανοποιημένο με, με αυτή τη συζήτηση. Η πρόεδρος. Ίσως μπορούμε να βελτιώσουμε τις μελλοντικέ ε, αυτές συναντήσεις. Θα δούμε. Μαρία, ναι. Εγώ Είχα μια συνάντηση μόλις με το Πανεφρικανικό Κοινοβούλιο που το συζητήσαμε και το θέμα αυτό για τη συμφωνία μετά το Κοτονού και ο πρέσβης Αφρικανικής Ένωσης που ήταν παρόνα ξέφρασε την απογοήτευσή του ε, κατά κάποιο τρόπο για το ότι η Αφρικανική Ένωση έχει ένα συμβουλευτικό λίγο πολύ ρόλο. Δηλαδή τίποτα από όσα άλλα δεν είναι δεσμευτικά. Και τώρα προσπαθεί να βρει, να εξασφαλίσει, αν θέλει ένα καλύτερο ρόλο για την Αφρικανική Ένωση σε όλε αυτέ τι διαπραγματεύσει. την επόμενη φορά, ε, ελπίζω πάντω να έχουμε περισσότερη ενημέρωση. Ίσως λοιπόν την επόμενη φορά μπορούμε να συζητήσουμε και το ρόλο τη Αφρικανική Ένωση, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων αυτών, διότι είναι κάπω δύσκολα τα πράγματα για την Αφρική. 48 χώρε ΑΚΕ, Βόρεια που δεν είναι στι χώρε ΑΚΕ, αλλά είναι στην Αφρικανική Ένωση και είναι δύσκολο ο ρόλος. Δεν έχουν και κοινή θέση ουσιαστικά για την Ολύπηρο. Και ήταν ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε ο Πρέσβης. Πραγματικά εξέφρασε την απογοήτευσή του. Ξεκάθαρα απογοητεύσει για την κατάσταση. Πρόεδρος, πράγματι. Εντό Αφρική υπάρχουν διαφορετικέ απόψει. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει στην Αφρικανική Ένωση ένα πιο μείζωνα ρόλο. Πρέπει τα αφρικανικά κράτη να καταλήξουν. Αυτό το σημείο ήταν προ ενημέρωση βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρξουν εξελίξει που θα απαιτήσουν μια νέα συνεδρίαση τη ομάδα παρακολούθηση πριν τι εκλογέ. Αυτό που είπε ο Επίτροπο Μίμητσα για τι διαπραγματεύσει μαρτιο Μάρτιο, Φεβρουάριο-Μάρτιο. Έχουμε μια συνάντηση επιτροπή μέχρι τι εκλογέ. Τέλο πάντων, θα παρακολουθούμε τα πράγματα και αν προκύψει κάτι νέο, θα το συζητήσουμε πριν τις εκλογές, αν όχι θα εκλειφθεί το επόμενο κοινοβούλιο, η νέα επιτροπή μας. Εσάς ευχαριστώ λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι. Μπορώ λοιπόν να κλείσω τη σημερινή συνεδρίαση νωρίτερα ε, για αλλαγή. Καλό είναι αυτό. Έξι ώρα λοιπόν λίγουμε. Αύριο 9 το πρωί η συνεδρία των συντονιστών. Και οι υπόλοιποι έχετε άλλη μια ωρίτσα ξεκούρασης ε, πριν έρθετε στις 10 για τις ψηφοφορίες. 10 για τις ψηφοφορίες. Καλό βράδυ.